Καλησπέρα. Πρώτο σημείο, η έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης. Θα πρέπει να ξεκινήσει η συνεδρίασή μας ε, με την αναφορά του κυρίου Βίλαντ για την αποστολή στην Αυστρία. Επίσης έχει μοιραστεί και ένα κείμενο προφορικής ερώτησης. για να παρουσιαστεί και στη διάσκεψη των Προέδρων ε, και να μπει στην ημερήσια διάταξη μία των επομένων ε, ολομελιών. Μετά ο, κύ... Κυρία Μέγερ, κύριος Μέγερ θα πρέπει να ξεκινήσουμε την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών. Μετά η κυρία Τουργάης θα κάνει την παρουσίασή της και θα έχουμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα είναι παρόντες στην αίθουσα ή αναφέροντες για τις αναφορές αριθμός 8 για ε, μία χωματερή στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία στη Γαλλία και μία στην Πολωνία. Α, ο Ντέβιτ Λόου μου είπε ότι υπάρχει μία διαφορά. Δεν θα έχουμε τον ε, υπογράφοντα την αναφορά στο 10. Ενώ θα είναι παρόν ο υπογράφων την 13 για τις ε, υποδομές ε, στην Ελλάδα. Τώρα για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου κυρία Όκεν θα μιλήσει και για αύριο το πρωί θα έχουμε τους αναφέροντες των σημείων 17 δεν θα είναι παρόν ο αναφέρον, ο κύριος Κρόιτσμαν θα είναι παρόν, ο εισηγητής της ΣΥΝΚΟ. Δυστυχώς οι αναφέροντες δεν δέχτηκαν την πρόσκληση την τελευταία στιγμή. Και θα είναι παρόν ένας εκπρόσωπος της ε, Αυστραλιανής Πρεσβείας Παρατιενώση. Μετά θα έχουμε τους αναφέροντες του 19 για, τις, για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Μετά στην 20 για τη Σόρια και την Ουμάνθια στην Ισπανία. Μετά για την 22 σχετικά με το αεροδρόμιο του Φουεντεράμπια και την 25 για την κτηνοτροφία στο Κίλκενι, στην Ιρλανδία. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Πάμε στο σημείο 2, έγκριση των πρακτικών της 24ης-25ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου. Έχουν μοιραστεί τα πρακτικά και αν δεν έχετε σχόλια εγκρίνονται. Εγκρίθηκαν λοιπόν. Πριν από μια εβδομάδα μοιράστηκε ο κατάλογος των αναφορών που προτείνουμε να κλείσουμε και αυτό λόγω έλλειψης απαντήσεων και αυτόν επίσης που πρέπει να ξανανοίξουμε λόγω των επιπλέον πληροφοριών που λάβαμε. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία παρατήρηση, οπότε αυτές οι συστάσεις εγκρίνονται. Σας πληροφορώ ότι η γραμματεία εργάζεται για την σύνταξη ενός πληροφορικού δελτίου, ένα newsletter, και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να συνεισφέρετε στην σύνταξη. Θα τα πούμε όμως και στους συντονιστές αυτά. Αν δεν έχετε άλλες τοποθετήσεις, πάμε στο 5. Κοίταζα, κοίταζα γύρω μου όντως είναι απόνο ο συνάδελφος Βίλαντ. Οπότε πάμε με το σημείο 6, αν ο αντιπρόεδρος Μέγερ ε, είναι διαθέσιμος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε στη φάση των πρώτων ανταλλαγών, στην πρώτη φάση των ανταλλαγών απόψεων και μπορούμε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε πιο αναλυτικά σε αυτή τη δεύτερη φάση. Έχουμε εμεί τους αριθμούς ε, για όλες τις εκθέσεις που συντάσσουμε και φυσικά έχουμε το περιγραφικό μέρος ε, για τις ανοιχτές, κλειστές ή ε, εκκρεμείς αναφορές, πώς μας ήρθανε, με ποιον τρόπο, άμεσα οι αναφέροντες ή κατέθεσαν την αναφορά μέσω ίντερνετ. Θα γίνει δηλαδή μια περιγραφή όσο το δυνατόν πιο πλήρης. Οι αναφορές ήταν 1646 για το 2010. Είχαμε μια ελαφρή διαφορά με το 2009. Ολοκληρώσαμε το 58,3%, παρέμειναν ανοιχτές το 21,5% και 3% αρχιοθετήθηκε. Από τις 1646 αναφορές οι περισσότερες ήρθαν μέσω της ιστοσελίδας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αντίστοιχο ποσοστό με το 2009 και μετά είχαμε τις μέσω ταχυδρομείου 35,6%. ανάλογα με τις χώρες έχει γίνει μια αλλαγή. 15,4% προηγείται η Ισπανία και ξεπερνάει τη Γερμανία. Αυτό θυμίζει ποδόσφαιρο αλλά δεν είναι. Μετά έχουμε Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα, Πολωνία, Γαλλία. Η Ιταλία ήταν πρώτη και μετά είχαμε την Ισπανία. Άλλαξαν λοιπόν οι αναφέροντες. Για τις γλώσσες. Οι αναφορές που λάβαμε ήταν 28,8% γερμανικά, 16,6% αγγλικά, 11,8% τα ιταλικά, 15% και κάτι τα ισπανικά, ίδια σειρά με το 2009. Πρώτο θέμα το περιβάλλον. περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ε, διατήρηση, προστασία του περιβάλλοντος και μετά θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη. Αυτού του είδους οι αναφορές υπερίσχυσαν την τελευταία χρόνια. Θα έπρεπε να συντάξουμε μία έκθεση με αυτές τις γενικές ε, θεωρήσεις και μετά με πιο συγκεκριμένες ε, θέσεις αξιολόγησης αξιολόγηση θετική ή αρνητική, λάθη που διαπιστώσαμε το 2010 και που θα μπορούσαμε να διορθώσουμε. Πρέπει να επιμείνουμε στο σημαντικό ρόλο αυτής της Επιτροπής, ε, προστασία της άσκησης, του δικαιώματος υποβολής αναφοράς από τους Ευρωπαίους πολίτες, Πρέπει επίσης να καταγράψουμε τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίσαμε στην Επιτροπή Αναφορών και αυτό να το δώσουμε ως παράδειγμα και μετά τις αποστολές τις οποίες ε, κάναμε το 2010 στην Καμπανία, στην Χουέλβα, στην Αυστρία και πρέπει να πούμε να τονίσουμε τον καλό συντονισμό αυτής της Επιτροπής ε, με τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Θα έπρεπε μετά από αυτήν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων να αρχίσετε και εσείς να λέτε τη γνώμη σας ε, για το αξιολογικό μέρος ε, και η κάθε ομάδα θα έπρεπε να αρχίσει να ορίζει τη θέση της και να έχει υπόψη της και το χρονοδιάγραμμα. Ένα, 1η Μαΐου θα έχετε το τελικό κείμενο του σχεδίου έκθεσης, θα φύγει για την μετάφραση. 12 Μαΐου θα έχει μεταφραστεί. Θα το παρουσιάσουμε 23 Μαΐου στην Επιτροπή Αναφορών. Μέχρι 30 Μαΐου για την κατάθεση τροπολογιών και θα ψηφίσουμε 14 Ιουνίου στην Επιτροπή και θα περάσει από την Ολομέλεια τον Ιούλιο. Λέω λοιπόν από σήμερα να ξεκινήσουμε την ανταλλαγή απόψεων, να πει η κάθε ομάδα τη γνώμη της και να αρχίσουμε να συζητάμε για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο συλλογική έκφραση στην έκθεση αυτής της Επιτροπής. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μέγερ για τη δουλειά του. Ζητώ από τους συναδέλφους, αν θέλουν να ξεκινήσουν τη συζήτηση. Θέλει κανείς το λόγο. Ο συνάδελφος Γιάρ. Μία σύντομη παρατήρηση. Ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί Εάν θέλετε, με αυτή την έκθεση κάνουμε και μια διαφήμιση της Επιτροπής μας. Είναι σημαντικό να καταγράφουμε τη δουλειά μας και όσον αφορά τις προτάσεις θα θεωρούσα λογικό να παρακαλέσω τον εισηγητή να γίνει μια συζήτηση με τους κοιοδησίγητες, ε, τον εκπρόσωπο της κάθε ομάδας και τότε θα έχουμε αυτή την ε, έτσι, πρώτη συμφωνία γιατί θέλω να το πω εγώ δεν θεωρώ πως είναι τόσο έτσι επίμαχη αυτή η έκθεση από πλευράς ε, πολιτικής και υπάρχει έτσι ο κίνδυνος να περάσει στον τούκο. Οπότε για εμένα πάντα είναι ένα ερώτημα σημαντικό γιατί πράγμα είμαστε υπεύθυνοι και γιατί όχι. γιατί βεβαίως έχουμε αιτήματα που φορούν τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας, ε, το δεχόμαστε, αλλά μετά βλέπουμε πως νομικά δεν είμαστε ακριβώς υπεύθυνοι. Και το δεύτερο ερώτημα για μένα είναι σχεδόν σημαντικότερο. Έχουμε αιτήσει για τις οποίες είμαστε αρμόδιοι, αλλά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί οι οδηγίες είναι αντίθετες και λέμε ως Επιτροπή η κατάσταση ε, συμβιβάζεται. Οπότε θα έπρεπε να βρούμε κάποια σύνδεση αν θέλετε ότι δεν ε, είμαστε εδώ πέρα μόνο για να χάσουμε τον κόσμο και να λέμε σας καταλαβαίνουμε αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αλλά θα πρέπει να δίνουμε και κάποια ερεθίσματα αν θεωρούμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει κάποιον ε, κανονισμό. Μπορούμε λοιπόν η οδηγία να δώσουμε στην Αναλόγη Επιτροπή ε, κάποιο ερέθισμα για να αδειάσει, να αλλάξει με σχόλια. ο κανονισμός. Ε, δεν έχω διαβάσει εδώ πέρα συγκεκριμένα το, το κείμενο, αλλά θα πρέπει να γίνουμε ένα σύνδεσμος μεταξύ των πολιτών και των αρμοδίων επιτροπών. Και ξανά η παράκληση να οργανωθεί μια συζήτηση για να συζητήσουμε το θέμα λεπτομερώς. Για να εγκριθεί και μετά νομίζω θα εγκριθεί και σχεδόν ομοφωνία. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Κάποια σχόλια έχω. Απευθυνόμενοι προς τον Πίτερ και στα όσα μας είπε. Διαφωνώ σχετικά με το ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα για το θέμα αυτό. Ε, είχαμε καλή πλειοψηφία στην πρώτερη θητεία του Κοινοβουλίου ψήφισε την έκθεσή μου για την Ισπανία. Την πέρασε, ήταν κατά το ΕΛΚΑ, αλλά ήταν μεγάλη πλειοψηφία που την ψήφισε. Και είχα μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα που υπερψήφισε τον Ουγγρικό νόμο για τα μέσα ενημέρωση. Δεν ενδείκνεται να λέμε ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου απέτυχε. Δεν μπορεί να το πει αυτό η πλειοψηφία εδώ. Έχουμε την αρμοδιότητα όπως περιγράφεται στο άρθρο 7. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να συζητήσουμε τις αρμοδιότητες και να πούμε ότι ένα από τα ζητήματα για ανθρώπινα δικαιώματα και κατά πόσο εφαρμόζονται, μπορούν να εφαρμοστούν οι ατάξεις ανθρώπινα δικαιώματα της εργασίας της Επιτροπής. Τα είδαμε τα θέματα, χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση, διότι έχουμε πολλές υποθέσεις με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωση στη Ρουμανία, και στην έκθεσή μου για την Ισπανία, τον Ισπανικό νόμο, τίθεται αυτά τα θέματα. Βίλι Μάιερ, θα ήθελα η έκθεσή μας να είναι πιο συγκεκριμένη από ό,τι πέρσι. Είναι εύκολο όλοι να είναι πολύ γενικόλογοι, με επικεφαλίδες ούτως υπήν. Χρειάζεται να φέρουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι κάνουμε για να δούμε τι προβλήματα αντιμετωπίσαμε για τη σύνταξη της εκθέσεως. Και σχετικά με αυτό να πω ότι στην έκθεσή σου θα έπρεπε να αναφέρεις αυτό που περάσαμε πριν από τις εκλογές το 2009 όπου ζητήσαμε από αυτή την Επιτροπή να επισημοποιηθεί περισσότερο. Έχει και, υπάρχει και πρόβλημα με την ονομασία. Κανείς στη χώρα μου δεν ξέρει τι ακριβώς κάνει αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να αναφερόμαστε και στην αναφορά των πολιτών. Θα είναι πιο εύκολο να το καταλάβουν οι λαοί εκείνοι που δεν έχουν ε, επιτροπή αναφορών στο Κοινοβούλιο. Κανεί στις σκανδιναβικέ χώρες δεν έχει την παραμικρή ιδέα σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής μας. Το όνομα είναι κενό γράμμα, δεν καταλαβαίνω τίποτα η ονομασία. Και στη Σουηδία ισχύει το ίδιο. Αυτό που δεν πέτυχε η προηγούμενη έκθεση, ο David Hammerstein την ετοίμασε νομίζω, που εγκρίθηκε. Αυτά δεν πέρασαν. Αυτή η έκθεση θεωρώ ότι είναι πολιτικό εργαλείο. Θα έπρεπε να είναι πολιτικό εργαλείο με το οποίο μπορούμε να ενημερώνουμε ακόμα και τους συναδέλφους μας σχετικά με αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλοσύνη σας, διότι είναι δική σας έκθεση και σύμφωνα με το άρθρο 282 υποβάλλεται έκθεση στην Ολομέλειά σας. Θα ήθελα να αναφερθώ όμω σε ένα-δύο πράγματα που έφυξε η κυρία Άουκεν και ο κ. Μάιερ. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι από καιρού καιρών πρέπει να θυμόμαστε ότι και το Κοινοβούλιο είναι νομοθετική αρχή και κάποια ε, στοιχεία πρέπει, ε, που αναφέρονται, πρέπει να τίθενται στην προσοχή της Αρμόνης Επιτροπής. Για το έτος 2010 είχατε πριζωθεί περισσότερο, μπορώ να το πω, στις βασικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. συμμετείχατε ακόμα και σε νομοθετικό θέμα που ήταν η πρωτοβουλία των πολιτών. Και αυτή η μεγαλύτερη εμπλοκή σας στις εργασίες του Κοινοβουλίου μετά τη Λισαβόνα, στα πλαίσια της θέσπισης νομοθεσίας, ε, είναι κάτι που πρέπει να τονιστεί και να υπογραμμιστεί. Και η κυρία Άουκεν είπε ότι πρέπει να δείξουμε καλύτερα ε, το τι γίνεται στην Επιτροπή μας, τι έργο παράγουμε και θεωρώ που είμαι φιλικός παρατηρητής από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αν συνδέεστε με τις βασικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις νομοθετικές του δραστηριότητες, αυτό είναι μια εύκολη προσέγγιση, είναι ένας εύκολος δρόμος για να πετύχετε αυτό που θέλετε. Ευχαριστώ. Και εγώ εκφράζω και τη δική μου φιλία, ανταλλάσσουμε συναισθήματα φιλία προ τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω τελικά να υλοποιηθούν και σε ένα πτυσίασμα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Επιτροπή μα. Δέχομαι λοιπόν προτάσεις, τις προτάσεις και τις σκέψεις που εξέφρασε ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι άλλοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα καλούσα λοιπόν τους υπευθύνους των ομάδων να μας πούν ποιοι θα είναι οι σκιώδεις συζητητές, ε, ούτως ώστε και στους συζητητές να δώσουμε τη δυνατότητα, στον συζητητή να δώσουν τη δυνατότητα να ε, προβούν στην ανταλλαγή απόψεων όπως πρότεινε και ο συνάδελφος Γιάρ. Κύριος Βίλαντ έχει έρθει, στρέφομαι στο σημείο 5 δίνοντάς του το λόγο για την, έκθεση, για την παρουσίασή του, την εισαγωγική για την αποστολή στην ε, Αυστρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το ότι αναβάλατε το θέμα για κάνα δύο λεπτάκια. Είχα και άλλη μία έκθεση για τις χώρες ΑΚΕ, που δεν είναι Αυστρίας Καραϊβικής Ειρηνικού, αλλά Αφρικής Καραϊβικής Ειρηνικού. Εν πάση περιπτώσει, έδωσα μια... Σας είπα τα της έκθεσης ε, της κυρίας Μπέργκερ Ξέρετε πως ε, τα συμπεράσματά μας τα συμπεράσματά μας είναι σαφή και βεβαίως οι δύο συνάδελφοι συμφώνησαν με το κείμενο αυτό Θεωρούμε λοιπόν πως ε, θέλουμε σαφείς πληροφορίες από την ε, Κομισιόν. Νομίζω έχετε όλοι το σχέδιο κειμένου και υπάρχει ένα προφορικό ερώτημα προς την Επιτροπή το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από την Κομισιόν για να προγραμματίσουμε τα επόμενα βήματά μας. Κατά βάση δηλαδή έχουμε το ερώτημα πόσο, σε ποιο βαθμό μπορούμε να ρυθμίσουμε τέτοια έργα τοπικά, χρονικά ή με άλλο τρόπο όσον αφορά το διαχωρισμό τους και εξ άντε και εξ πόστο αναλόγως στην ε, περίπτωση υπάρχει εδώ πέρα κάποιος ο οποίος έχει υποβάλει ένα σχετικό αίτημα. Και το δεύτερο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα προσωπικά ζήτημα είναι σε ποιο βαθμό οι πίστες του σκι που δημιουργούνται χωρίς να αλλάξει το έδαφος θα πρέπει να μείνουν εκτός ε, της ε, αρμοδιότητας ε, της περίπτωσης αυτής, γιατί κατά την άποψή μου δεν έχουν κάνει κανένα ουσιαστικό λάθος εκεί πέρα οι τοπικές αρχές, αλλά εάν αφήνει τελείως τις, λίστες, τις πίστες ε, του και ένα κράτος μέλος εκτός, δεν ξέρω εάν πρόκειται περί σωστής εφαρμογής της ανάλογης οδηγίας έχω τις αμφιβολίες μου, εξού και η προφορική αυτή ερώτηση. Και ανάλογα με την απάντηση που θα λάβουμε, θα μπορέσουμε να κρίνουμε εάν και τι πρέπει να κάνει παραπέρα η Κομισιόν. Εάν δηλαδή θα αρκέσουν οι διευκρινήσεις, εάν θα πρέπει να καταφύγουμε σε άλλα πιο σοβαρά μέσα. Ευχαριστώ κύριε Βίλαντ. Θέλει το λόγο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ωραία μουσική ακούμε εδώ. Λοιπόν, όσον αφορά τις νομικές πτυχές, Γνωρίζουμε ότι η οδηγία για την αξιολόγηση που αφήνει μεγάλη ευελιξία στα κάτι μελη Αυτή η ευελιξία όμως δεν είναι απεριοριστή. Όταν έγινε αυτή η αναφορά, η Αυστρία παραβίαζε κατάφορα την οδηγία, η Αυστρία άλλαξε την ομοθεσία της και τώρα συμμορφούται με αυτήν. Η συμμόρφωση είναι επί χάρτου τέλεια, αλλά παραμένει ακόμα μεγάλο επίπεδο, μεγάλο περιθώριο ευελιξία για του επιτόπου εφαρμόζονται στην οδηγία. Χρειάζεται λοιπόν προβλεψιμότητα, σαφήνεια όχι μόνο για προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για του επιχειρηματίε να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βοήθεια τη Επιτροπής σα είναι να δίνουμε περισσότερε οδηγίε ε, και πώ πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες. Έχουμε ένα εγχειρίδιο εδώ σχετικά με την απόφαση με την οδηγία, με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το κείμενο βρίσκεται στο σελίδα. Είναι ευφυή η ιδέα του κ. Βίλαντ, διότι επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν απαντά στο ερώτημα ω σώμα, να παρέχει και άλλε οδηγίε όσον αφορά το τι είναι εφικτό και τι είναι ανέφικτο σύμφωνα με την οδηγία. Επίση, έτσι εξασφαλάζεται ισότιμη αντιμετώπιση όλων των κρατών μελών και αυτό είναι σημαντικό παράγοντα για τον Επίτροπό μου και επίση συνδέεται αυτό και με την αναθεώρηση τη οδηγία. Καταρχά, λοιπόν, καλωσορίζουμε την αποστολή αυτή που έλαβε χώρα, την επίσκεψη στην Αυστρία και η προσέγγιση που ακολουθείται από την Επιτροπή σα και προτείνεται από τον κύριο Βίλαντ είναι πολύ καλή. Επί τη βάση μια υποθέσεως που νομικώ έχει επιληθεί, μπορούμε να βελτιώσουμε περισσότερο τη διαφάνεια και την προβλησιμότητα των κανόνων. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ συνάδελφε Βίλαντ. Να ακούσουμε μήπως κάποιος από τους συναδέλφους θέλει να τοποθετηθεί και μετά να πάρετε εσείς το λόγο. Ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Βίλαντ. Δύο πράγματα. Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το αρχικό κείμενο, αν είναι αυτό ή όχι. Ε, στο τέλος αυτού του κειμένου έχει κάτι παύλες, στην τέταρτη παύλα στα γερμανικά μιλάτε εδώ πέρα για νομολογία. Αλλά εννοούμε την νομοθεσία. Και για την νομική μορφή, δηλαδή αν κάποιος ιδρύσει δύο εταιρείες, ε, εν πάση περιπτώσει πρέπει να διορθωθεί η γερμανική μετάφραση. Ευχαριστώ λοιπόν την ε, Κομισιόν για αυτά τα οποία είπε, τα οποία δεν μας βοηθάνε βέβαια και πολύ. Να πω λίγο τι εννοώ. Και εγώ θέλω ευελιξία, αλλά ως ποιο βαθμό μπορούν να αποφασίζουν με ευελιξία οι τοπικές ε, αρχές ε, ε, και αν προσφέρει αν θέλετε κάποιο χώρο δημιουργικότητας. Υπάρχει μια διαφορά εδώ πέρα. Δηλαδή, αν έχουμε μία έκταση 100 εκταρίων και έχουμε ε, δύο lift ε, του σκι, είναι προφανές πως δεν μιλάμε για ολόκληρη αυτή την έκταση η οποία καλύπτεται, αλλά από την άλλη τον χειμώνα κατά τη διάρκεια της ημέρας προφανώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πανίδα αυτή η έκταση. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποιος συντελεστή εάν θέλετε. Εάν φωτίζω παραδείγματο χάρη τη νύχτα, την πίστα ή εάν κάθε νύχτα ε, ρίχνουμε τεχνητό χιόνι, είναι τελείως διαφορετικός ο συντελεστή ε, της ε, πανίδας. Και αν μετά εξοπλίζουμε, εξοπλίζουμε το lift και βάζουμε διπλάσιο αριθμό καθισμάτων και έρχονται πολύ περισσότεροι άνθρωποι επάνω και αυτό διαφέρει. Αλλά βλέπετε τις νέες δυνατότητες ε, που υπάρχουν και για το σκι με το carving ή να πηγαίνει κάποιος ο οποίος δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε πολύ βαθύ χιόνι ή τους λεγόμενους, ας το πούμε, ελαφρεπιβάτε εν πάση περιπτώσει, κάποιο ο οποίος βγαίνει εκτός της ε, πίστας. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη όταν κάνουμε ε, μελέτη περιβαλλοντικών ε, αντικτύπων και να δούμε τουλάχιστον πώς μπορεί να εμποδιστεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, θα μπορούσατε να τα λάβετε αυτά υπόψη στην απάντησή σας ήδη. Ε, Νομίζω ότι όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στις ερωτήσεις που υποβάλλουμε στην Κομισιόν και στην προφορική ερώτηση. Δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις. Ζητώ από την Επιτροπή να ψηφίσουμε την έκθεση Βίλαντ και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνεται ομόφωνα. Όπως επίσης και η προφορική ερώτηση που μοιράστηκε στην αρχή των εργασιών. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα η ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Βίλαντ. Σημείο 7. Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων. Ο Αντιπρόεδρος Ιτουργάης έχει το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Κυρία Πρόεδρε, όπως και στο σημείο 6 του φίλου και συναδέλφου Μπίλι Μέιερ, πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων. Εμείς δεν μπορούμε, δεν έχουμε βέβαια μπροστά μας κανένα κείμενο, αλλά θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να σας πληροφορήσω σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό. Έχουμε πολλές αναφορές ακόμη και στη σημερινή ημερήσια διάταξη σχετικά με απόβλητα και περιβάλλον. Είναι ένα θέμα καυτό, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Όπως ε, θα γνωρίζετε σήμερα στους συντονιστές ε, στο πέρας αυτής της συνεδρίασης θα συζητήσουμε υπό ποιους όρους θα συνταχθεί η εξωτερική έκθεση που ανέθεσε η Επιτροπή Αναφορών για τη διαχείριση των αποβλήτων ανά την Ευρώπη. Και θα ήθελα να κάνω σχετικά μερικές θεωρήσεις. Αυτή τη μελέτη τη ζητήσαμε εμείς οι συντονιστές των διαφόρων ομάδων. Διότι αν δεν έχουμε τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης δεν μπορούμε να συντάξουμε κανένα προσχέδιο έκθεσης. Η γραμματεία βέβαια με πληροφόρησε ότι σε τρεις μήνες θα ολοκληρωθεί η μελέτη. Κυρία Πρόεδρε, πάνω κάτω τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Δηλαδή η πρώτη παρουσίαση της έκθεσης πρέπει να γίνει μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Όμως μέχρι να έρθει η έκθεση πρέπει να σας πω ότι δεν πρόκειται να σταματήσω εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ε, γραμματεία για την ε, βοήθειά τους. Και σε αυτήν την ε, παρένθεση που θα ανοίξει τώρα μέχρι να έρθει η εξωτερική έκθεση θα συλλέξω όλα τα σχετικά τεκμήρια και τις στατιστικές για τη διαχείριση των αποβλήτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συντάξω έναν κατάλογο για όλων των αναφορών που εξετάσαμε σχετικά με τα απόβλητα, όπως επίσης και τις οδηγίες που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση όπως επίσης και μία ανάλυση των προβλημάτων για την εφαρμογή της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα πόβλητα. Όλα αυτά θα, είναι θα αποτελέσουν τα βασικά σημεία, τον βασικό κορμό της έκθεσης και όταν θα τα έχουμε όλα αυτά θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία με τους και όδης εισηγητές γύρω από το θέμα. Αυτή είναι η διαφορά της δικής μου έκθεσης με την έκθεση του κυρίου Μέγερ που θα έρθει έγκαιρα. Αλλά εγώ θα πρέπει να περιμένω την έκθεση των ε, εξωτερικών εμπειρογνωμών. Βέβαια εν αναμονή θα προχωρούμε με περιορισμένα βήματα μέχρι να έρθει η έκθεση και μεταφρασμένη στις διάφορες γλώσσες. Στο μεταξύ εγώ είμαι στη διάθεση των συναδέλφων αν κάποιος θέλει να με ρωτήσει κάτι. Ευχαριστώ. Κύριε Τουργάη. θέλει κανείς το λόγο. Η συνάδελφος Μέρκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφε. Πάρα πολλές αναφορές παρελήφθησαν από εμά για όλα τα είδη των αποβλήτων. Θα κάνετε κάποια διαφοροποίηση, όπως αναφέρεται στο πρώτο εκεί κείμενο για τα θέματα αποβλήτων, θα εστιαστείτε συγκεκριμένα θέματα περί αποβλήτων ή μη γενική επισκόπηση θα κάνετε. Το ερώτημά μου, η μελέτη θα υπάρχει ελεπικάλυψη με την έκθεση ή θα συμπεριλάβατε εξ ολοκλήρου τη μελέτη στην έκθεσή σας. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει υποπέσει την προσοχή Τη επιτροπή, αλλά πρόσφατα Το Ιανουάριο ο επίτροπο Πατότσνικ παρουσίασε την πλήρη επισκόπηση των θεμάτων αυτών, των αποβλήτων και τη διαχειρίσεως αυτών και αφορά αυτό την εφαρμογή των, ε, του κανονισμού περί αποβλήτων σε όλα τα κράτη-μέλη. Με σαφή στατιστικά στοιχεία για τι επιδόσει. Νομίζω λοιπόν ότι εν μέρη αυτό που θέλει να πετύχει η μελέτη έχει επιτευχθεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραμένει λοιπόν το ερώτημα. Τι θα κάνουμε όσον αφορά την έκθεση. Πώς θα ανοίξει το δρόμο αυτή για τους αναφέροντες που μας απευθύνθησαν κατά το παρελθόν. Μπορούμε να παρουσιάσουμε μια παρηγοριά, να δώσουμε μια παρηγοριά, να τους δώσουμε μια κάποια λύση για αυτά τα θέματα. Θα προτείνεται ένα κάποιο ε, τύπο συγκεκριμένη προσέγγιση, θα πηγαίνουμε πάντα για μια αποστολή επιτόπια, θα έχετε συγκεκριμένη διαδικασία για τα θέματα αποβλήτων, γιατί φοβούμαι ότι στο μέλλον τα θέματα αυτά θα γίνουν ακόμα πιο αριθμά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μέρκη. θέλει κανείς άλλο το λόγο. Μπορείτε να μας πείτε πότε θα γίνει η επόμενη ανταλλαγή των απόψεων, παρακαλώ. Nessun άλλο la parola. Κανείς άλλος δεν θέλει το λόγο. Η κυρία Όκεν. Ναι. Συγγνώμη, δεν ήξερα το, το θέμα. Έπρεπε, έπρεπε να το έχω δει γιατί είναι θέμα περιβάλλοντος, το ξέρω. Βεβαίως μπορούμε να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Να δούμε και με τη γύρω τι, τι συμβαίνει. Βεβαίω θα το κάνετε αυτό γιατί όλοι ενδιαφερόμαστε για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας εδώ πέρα και οπωσδήποτε το θέμα, τα θέματα των αποβλήτων ε, θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια. Ε, ακούμε ε, τι γίνεται ε, όταν μαθαίνει ο κόσμος πως μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να έρθει σε μας, οπωσδήποτε τότε θα, θα αυξηθεί ο όγκος. Οπότε συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε και ελπίζω να έχουμε επικοδομητική εργασία. Ε, Κανείς άλλος. Καλό τους συντονιστές να μας ορίσουν ποιοι είναι οι σκεώδεις εισηγητές και να μπορέσουμε να έχουμε μία πλουραλιστική αντιπαράθεση γύρω από τις εργασίες μας. Και θα προχωρήσουν παράλληλα με την μελέτη. Θα κοιτάξουμε δε να υλοποιήσουμε όλα αυτά το συντομότερο. <coughs> Συνάδελφε Μέρκης, εγώ σήμερα δεν είμαι σε θέση να δώσω ημερομηνία για το επόμενο ραντεβού. Θα το δούμε, θα το εξετάσουμε και με τους ε, εισηγητές, ε, τους κοιόδης εισηγητές και τον εισηγητή. Ο συνάδελφος σου Τουργάης ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και κυρίως την συνάδελφο την κυρία Μέρκης για να της απαντήσω στις ερωτήσεις. Για το θέμα της ανταλλαγής απόψεων, εγώ βρίσκομαι σε μια κατάσταση αδιεξόδους και, και θα έλεγα σε ένα stand-by δεν το ζήτησα εγώ να, να γίνει αυτή η εξωτερική έκθεση. Όλες οι ομάδες το είχαν ζητήσει. Θα πρέπει δηλαδή εμείς να περιμένουμε για να μπορέσουμε ε, να αντιδράσουμε εμπρόθεσμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέγατε αν θα υπάρξει επικάλυψη ή όχι. Αυτό εξαρτάται από την έκθεση την ίδια. Εσείς μου είπατε ότι ήδη είχατε υπόψη σας άλλες εκθέσεις. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι εκθέσεις εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες ε, και μας ενημερώνουν ε, είναι ευπρόσδεκτες. Δεν ξέρω αν εσείς θα είστε η σκιώδης εισηγήτρια της σοσιαλιστικής ομάδας ή ένας άλλος συνάδελφός σας. Και τότε μπορούμε να τα βρούμε από κοινού. Θα ήθελα να συνεχίσω. Έλεγα λοιπόν ότι θα έχετε την ευκαιρία να συνεργα... θα έχουμε μάλλον την ευκαιρία να συνεργαστούμε έτσι όπως ε, με, με τον τρόπο που λέγατε εσείς. Και εγώ αυτό το οποίο περιμένω με αγωνία είναι να μπορέσουμε να εργαστούμε από κοινού και να εξετάσουμε όλα εκείνα τα θέματα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξωτερική έκθεση. Συγγνώμη Αντιπρόεδρε, δεν το είχα καταλάβει ότι ήθελε το λόγο. Πάμε στο επόμενο σημείο. 944-2004 σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποναφέρουσα την κυρία Σέιλα Έλλης, η οποία βρίσκεται εδώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, είμαι Σέιλα Έλλης και ο Colin Wakefield από την ομάδα κάτι κατά της τοξικού τη τοξική τοποθεσία. Αυτή η χωματερή δηλητηριάζει το περιβάλλον και την περιοχή του Όκνεσπρίνη. Το υψηλότερο σημείο τη πόλη είναι λιγότερο από 200 μέτρα από, από επιχειρήσει, από σπίτια και μαγαζιά. Είναι, είναι πολύ κοντά στο, ε, στον υδροφόρο ορίζοντα και έχουν οι βράχοι που είναι κοντά στη χωματερή και ε, ε, έχουν αποστεθεροποιηθεί γιατί ανεβαίνει το νερό από κάτω. Και βορειοανατολικά έχουμε το σταθμό άντληση στα 1,5 χιλιόμετρα του νερού. Και η υπηρεσία περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου πέτρεψε να ανοίξει αυτή η χωματερή το 1996, ξέροντα ότι περνάει πάρα πολύ γρήγορα το νερό μέσα από το υπόγειο νερό και από τα βράχια και ότι λιγότερο από 150 μέρε χρειάζονται για να περάσει το νερό σε αυτή τη διαδρομή και θα έπρεπε ε, να σταματήσει αυτή η Το Σάντερλαντ ήθελε να, να ρίξει τα σκουπίδια και μπήκε στη ζώνη 3 ώστε ε, να επιτρέπονται όλα τα απόβλητα εκτός από τα επικίνδυνα. Από τη στιγμή που άνοιξε η χωματερία άρχισε να μολύνει το περιβάλλον και η υπηρεσία ε, αποβλήτων δεν έκανε τίποτα και επανεισυρμένα παραβιάστηκαν οι όροι της αδείας στείλαμε email, έχουν καταγραφεί και η υπηρεσία η αρμόδια παραδέχτηκε ότι μολυνότανε το υπόγειο είδωρ, αλλά αυτό παρέμενε μυστικό, τόσο ώστε να αποφευθούν πολιτικέ συνέπειε με το Σάντερλαντ. Εξακολουθεί να μολύνεται το υπόγειο νερό με πολλά εκατομμύρια λίτρα που σπαταλιώνται σε μια προσπάθεια να σταματήσει, ε, στο να μην φτάσει το νερό το μολυσμένο στο, στο δημόσιο, στο νερό που, από το οποίο πίνει το νερό και η υπηρεσία έδωσε το 2004 και 2006 χαλαρές άδειες εκ νέου που παραβιάζουν του κανόνε του ενδροφόρου έπρεπε να κλείσουν κάποιε τοποθετησίε, διότι ήταν ασταθέ το υπέδαφο και δεν τόσο ασταθέ το υπέδαφο που ανοίγουν τεράστιε χαραγματιέ και τρύπε. Αλλά ο κανονισμό αγνοήθηκε και η κατάσταση δημόσια που περιγράφεται από του γεωλόγου, από τη γεωλογική και έρευνε είπαν ότι ήταν το χειρότερο μέρο να έχει κανεί χωματερή. Παρ' όλα αυτά η υπηρεσία επέτρεψε 350 είδη τοξικών αποβλήτων να πάνε εκεί, επικίνδυνα χημικά και άλλα είδη αποβλήτων. Κακό σχεδιασμό και κατασκευή σημαίνει ότι λίγα πράγματα μπορούν να σταματήσουν τη μόλυνση. Το πλαστικό περνάει το υπέδαφος και δεν τελειώνει στο, στον άργυλο το υπέδαφος ε, και τελικά υπάρχει μεγάλη μόλυνση και τα, τα, δεν μπορεί να πάει πάνω από μισό μέτρο το νερό για να συγκρατηθεί πάει στο 0,45 0,45 και τελικά πλημμυρίζει το νερό και μολύνει όλο το υδροφόρο ορίζοντα και ποτέ δεν καλύφθηκε η χωματερή. Η υπηρεσία είπε επανειλημμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είχε καλυφθεί από το 2002. Η αλήθεια είναι ότι εξακολουθεί να παραμένει ακάλυπτη και κάποια μέρη και, ε, τελικά συσσωρεύονται σε βουνό ε, τα απόβλητα ε, και, και αέρια επίσης ξεφεύγουν από τη χωματερή. Ε, βρωμάει, έχουμε μύγες, έχουμε σκουλίκια ε, έχουμε σύννεφα σκόνης ε, μολυσμένης και η υπηρεσία όλο δικαιολογίες βρίσκει. Και λένε ότι δεν μπορούν να ελέγξουν επαρκώ, δεν έχουν τον εξοπλισμό που έχει χαλάσει και η αρμόδια υπηρεσία δεν κάνει τίποτα. Προσπαθεί την αμέλειά τη να την καλύψει προσλαμβάνοντα εταιρείε για, να για να εγκρίνουν τι εργασίε τη τοποθεσία. Ε, είναι ίδιες εταιρείε όμως που το κάνουν αυτές που αγοράζονται, που πληρώνονται από την υπηρεσία που βάζει τα απόβλητα. Είναι αντίθετη προσέγγιση ε, που ακολουθεί η ΜΠΕΦΑ. Λοιπόν, και όλα υπάρχει κάλυψη. Λοιπόν, απελπισμένα οι κάτοικοι της περιοχής εστράφησαν προς το Κοινοβούλιο και ζητούν βοήθεια. Και σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε σε αυτά που είχαμε να πούμε. Eh, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με τρεις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Η Κομισιόν δεν έχει εξουσίες να κάνει επιθεώρηση. Οι συνάδελφοι από την Αμερικανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος μπορούν να το κάνουν εμείς ε, δεν μπορούμε να το κάνουμε, γι' αυτό χαιρόμαστε ε, για το ότι μας δίνουν πληροφορίες ε, οι αναφέροντες. Και η κυρία Έλλης είναι πολύ καλή πάροχος πληροφοριών. Κατόπιν, μετά από αυτό το οποίο ακούστηκαν, πώς είναι δυνατόν ένας χώρος υγειονομικής χωματερής να πάει τόσο κοντά σε σπίτια και πάνω από τα υπόγεια ύδατα. αυτό είναι ένα πρόβλημα της οδηγίας υγειονομικής ταφής ε, απορριμμάτων. Η πρόταση της Κομισιόν ε, ξέρετε πως ε, από τα κράτη-μέλη και μάλλον και από το εν κράτος μέλος εξασθένησε πάρα πολύ στο Συμβούλιο. Κανονικά αυτή η συμπεριφορά βεβαίω είναι θέμα των τοπικών δικαστηρίων. Οι πολίτε θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να πάνε με χαμηλό κόστο στα δικαστήρια και να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Το θέμα με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πω είναι πολύ ακριβή πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικασία επί παραβάση ε, ει βάρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Οπότε, ε, ε, ανακεφαλαιώνοντας, δεν έχει η Κομισιόν δυνατότητε. Επιτόπια έρευνα, ε, έλλειψη της οδηγίας και όπως σας είπα πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Τώρα, για την άδεια. Η άδεια εκτάθηκε το 2004 και ισχύει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πιέσουμε τις Βρετανικές αρχές να εξασκήσουν τον ρόλο τους από πλευράς επιτήρησης ε, το καλύτερο δυνατόν. Και όπως λέει και η κυρία Έλλης, είναι δύσκολο αυτό να γίνει. Λαμβάνουμε τακτικές αναφορές από τις αρχές για κάθε πτυχή του ΧΙΤΑ. Πράγματι έχει καθυστερήσει το, η κάλυψη της κομματερής. Ε, μας έχουν υποσχεθεί οι Βρετανοί συνάδελφοι ότι θα το κάνουν, οι Βρετανικές αρχές. Τώρα σε μια έκθεση του τέλους Φεβρουαρίου μας είπαν πως λόγω των ε, χειμερινών συνθήκων δεν ήταν δυνατόν. Ελπίζουμε να γίνει ε, σύντομα ακόμα και με το λάθος είδος χιονιού που λένε στη Μεγάλη Βρετανία. Ε, παρακολουθούμε επίσης την εξαγωγή αερίου από την χωματερή. Τώρα για τη μόλυνση των υπογείων υδάτων δεν ξέρουμε αν αυτή ακριβώς η αιτία. Υπήρχε ένας προσωρινός δρόμος πρόσβασης που έχει ε, κλείσει τώρα, που μπορεί να είναι η πηγή της ε, μόλυνσης. Έγιναν κάποιες έρευνες, Βεβαίω ξέρω πω οι ετούντε έχουν κάποιε αμφιβολίε για αυτά τα οποία λέει η Υπηρεσία Περιβάλλοντο του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά μπορείτε να είστε σίγουροι πω ε, αυτά τα οποία υποσχέθηκαν θα τα κάνει η Υπηρεσία Περιβάλλοντο. Οπότε παρακολουθούμε στενά, ασκούμε πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή μα ε, δίνει τι εκθέσει τι οποίε υποσχέθηκε. Η κατάσταση επιτόπου μπορεί να είναι κάπω διαφορετική. Γι' αυτό ε, είμαστε σε επαφή με τους ε, αναφέροντες για να επαληθεύσουμε αυτά τα οποία μας λένε οι αρχές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Κύριο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να πω πρώτα απ' όλα πως δεν έχω τη φήμη κανενός έτσι, φανατικού πρασίνου και αναγνωρίζω. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ τους συναδέλφους που το επιβεβαιώνουν και αναγνωρίζω πως ε, είναι μια, ένα αναγκαίο κακό οι χωματερές. Είδα όμως, ε, συνάντησα τους αναφέροντες και τη δουλειά που έχουν κάνει και μου φαίνεται εκ πρώτης όψεως πως έχουν πραγματικά ουσιαστικά ε, παράπονα. Οι Βρετανικές αρχές δεν εκπλήρωσαν τις προϋποθέσεις που έθεσαν οι ίδιες και αυτό το οποίο με ενισχύει ιδιαίτερα είναι πως οι Βρετανικές αρχές, από ό,τι φαίνεται, εσκεμένα και κατά εξακολούθηση υπέκρυπταν τα γεγονότα, προσπαθούσαν να μειώσουν τους αναφέροντες και προσπαθούσαν να αγνοήσουν το πρόβλημα αντί να το λύσουν και έτσι οι συνθήκες ε, αντί να ε, λύσουν το πρόβλημα και να εκπληρωθούν οι όροι της αρχικής άδειας. Η Κομισιόν ε, προσεγγίζει το ζήτημα όπως περιέγραψε και φαίνεται πως παρακολουθεί στενά το τι συμβαίνει, αλλά θα ήθελα να προτείνω, κυρία Πρόεδρε, πως καλό θα ήταν για την Επιτροπή μας να απευθύνει μια επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της Βρετανίας, να εκφράσουμε την ανησυχία μας και για τις συνθήκες οι οποίες φαίνεται ότι επικρατούν και για το ότι δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς και εγκαίρως ε, στα παράπονα των πολιτών. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Κάλμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα η θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Έλμερ. Εκπροσωπώ την περιοχή αυτή, τη βορειοανατολική, όπου βρίσκεται αυτή η χωματερή. Δεν θα πω ότι είχα τη χαρά να επισκεφθώ την τοποθεσία, δεν ήταν τα πραγματικά χαρά. Οι αναφέροντες ε, έχουν απόλυτο δίκιο, επανειλημμένα πήγα εκεί και όλα τα στοιχεία που έδωσαν είναι αληθινά. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστες οι περιβαλλοντικές συνθήκες εκεί και δέχομαι ότι υπάρχει ανάγκη χωματάει σε κάποιε περιοχέ, αλλά η τοποθεσία που επελέγει αντεδείκνυται, είναι πολύ κοντά σε κατοικίε, πολύ κοντά σε ένα κεντρικό δρόμο και πολύ συχνά ο αέρα παίρνει τα σκουπίδια και βγαίνουν στο δρόμο. Αλλά το θέμα της παραβιάσεως του ευρωπαϊκού δικαίου έπρεπε να μας απασχολεί και ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επί σειρά ετών αναφέρθηκε για το θέμα αλλά Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου ως υπεύθυνο φορέας δεν έλαβε στα σοβαρά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αναφέροντες ήταν πολύ καλά, πολύ καλοί. Ε, επί σειρά ετών έκαναν εκστατείες για το θέμα, έκαναν ό,τι μπορούσαν. Ε, ακολούθησαν και την τοπική δημοκρατική διαδικασία και οι δύο που είναι εδώ εξελέγησαν ως τοπική σύμβουλη εκπροσωπώντας την περιοχή. Ε, τόσο μεγάλες ανησυχίες έχουν οι κάτοικοι αυτά τα θέματα. Υπάρχει ιστορικό παραπλάνησης όσον αφορά τι πληροφορίε που δίνει η υπηρεσία περιβάλλοντο. Μετά από πολλέ διαμαρτυρίε, οι καταγγελίε παραδέχθηκαν τελικά με δισταγμό ότι τα υπόγεια νερά έχουν μολυνθεί και μόλις τώρα πολύ διστακτικά θέλουν να ερευνήσουν τι κάνει ο αρμόδιος φορέας και υπάρχει το ενδεχόμενο δίωξη. Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια μαχών και καταγγελιών και δημαρτυριών από τους ντόπιου κατοίκους και από την ομάδα ενημέρωσης και αν δεν έκαναν τις προσπάθειες αυτές θα είχε αποσιωπηθεί το θέμα και η εταιρεία θα μπορούσε να συνεχίσει και να ρηπαίνει το περιβάλλον. Θα ήθελα να προσφέρω όλη μου την υποστήριξη και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να λάβει κάποια δράση κατά τι υπηρεσίε περιβάλλοντο του Ηνωμένου Βασιλείου για το συγκεκριμένο θέμα και το μεταξύ θα ήθελα να υποστηρίξω τι ανησυχίε του συναδέλφου και ελπίζω η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλουν επιστολή στι Βρετανικέ Αρχέ και να ζητήσουν πληροφορίε στη συγκεκριμένη υπόθεση. Κυρία Όκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κοιτάω εδώ πέρα τα έγγραφα για να δω εάν οι πολλοί αυτές ενδιαφέρουσες πληροφορίες ε, και το κόστος του να πάει υπόθεση στα... Ποιο είναι το, το κόστος να πάει μια υπόθεση στα δικαστήρια και δεν μπορούν να πάνε οι απλοί άνθρωποι. Γιατί, ξέρετε, ε, αν τα κάνουμε εμείς όλα αυτά θα, θα πεθάνουμε σε αυτήν την επιτροπή. Γιατί τα εθνικά δικαστήρια απομακρύνουν τον κόσμο. Και είναι ανησυχητικό αυτό, αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω λοιπόν τι, τι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, μπορούμε να το συζητήσουμε και στην ε, συνεδρία συντονιστών. report, when I blame people... Θυμάμαι και από την Ισπανική έκθεση που κατηγορούσε τον κόσμο ότι δεν πήγε στα, στα δικαστήρια. Γιατί οι υποθέσει ήταν προφανώ για δικαστήριο. Και με πετάξαν έξω. Γιατί ε, αγνοούσα, δεν ήξερα το, το πώ δουλεύει το σύστημα ήταν αδύνατο να, να πάνε στα δικαστήρια και εκεί για άλλους λόγους. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ξεκάθαρη περίπτωση αν, το κόστος είναι τέτοιο που λέτε. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το οποίο μας είπατε. Αυτά. Και, και εγώ εξεπλάγει μου το άκουσα. Δεν ζητάει κανένα άλλο λόγο. Όσοι είναι Γιάρ. Οφείλω να συγχαρώ τους αναφέροντες. Εάν δει κανεί την ιστορία, εδώ πέρα το ιστορικό, υποθέτω πως η στρατηγική των αρχών ήταν ε, κολυσιεργία. Από το 2004 παλεύεται μέχρι σήμερα, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και άφηναν τα παράμονα αναπάντητα και σου λέει θα λυθεί μόνο του το πρόβλημα. Οπότε συγχαρητήρια για το ότι επιμείνατε. Το δεύτερο, βλέπω εδώ πέρα πως πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι ε, και εμείς ε, είμαστε, είμαστε βοήθητοι και ε, δεν ξέρω να μας φύγει η Κομισιόν τι μπορούμε να κάνουμε. Στο σημείο 8 εδώ πέρα βλέπετε αναφέρεται από την Κομισιόν πως οι Βρετανικές αρχές δήλωσαν πως το ότι ε, δεν ε, είχε ε, δεν υπήρχε σωστή επίστρωση και σφράγιση και θα πρέπει το κομμάτι 2 προσωρινά να κλείσει όμως δηλαδή εδώ πέρα είναι θράσος η μόνιμη ε, σφράγιση δεν θα ήταν δυνατή λόγω των ε, συνθήκων. Δηλαδή, τι, αν δεν είναι δυνατή η σωστή, η ορθή σφράγιση και το ομολογούν αυτό οι αρχές, τι, μπορούμε να κάνουμε από εκεί και πέρα. Εντάξει, σωστό να απευθύνουμε μία επιστολή στις Βρετανικές αρχές και ρωτά και την Κομισιόν τι άλλο σκέφτεται να κάνει. Γιατί από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχουμε μαζική και πεσχεμένη παραβίαση του δικαίου του, του περιβάλλοντος. Άμα είναι να κάνουμε έτσι δεν χρειάζεται να φτιάχνουμε νόμους. Όταν διαπιστώνει δηλαδή η ίδια η αρχή πως ε, προφανώς ε, έχει κατασκευαστεί η χωματερή σε μέρος το οποίο δεν θα έπρεπε καν, τι, να κάνουμε από εκεί πέρα. Ευχαριστώ κύριε Γιάρ. Εγώ πιστεύω ότι είναι αρκετά σαφή η θέση των συναδέλφων σε αυτή την Επιτροπή. Πρόκειται για μία σαφή καταγγελία των διαφόρων συμπεριφορών, έτσι όπως προκύπτουν <coughs> στην εξέταση αυτής της αναφοράς. Πρόκειται για μία αναφορά του 2004, 7 χρόνια πέρασαν. Και αυτά τα 7 χρόνια μεσολάβησαν πολλές φάσεις συζήτησης και αντιπαράθεσης. Η Κομισιόν πολλές φορές επανέλαβε αμφιβολίες γύρω από το θέμα και εξέφρασε και τις ανησυχίες της για τη σοβαρότητα των ε, γεγονότων. Αλλά παρόλα αυτά μετά από 7 χρόνια βρισκόμαστε πάλι εδώ και συζητάμε για ένα ζήτημα το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε. Νομίζω, όπως είπε και ο συνάδελφος Γιάρ, ότι θα έπρεπε να γίνει και πάλι μία ανακοίνωση προς τις Βρετανικές αρχές. Και όπως έλεγε και ο κύριος Κάλαγαν, θα πρέπει να γίνει και μία ανακοίνωση στο Ιστιτούτο για το περιβάλλον. Αλλά επίσης ε, θα έλεγα ότι πρέπει να ζητήσουμε και από την Κομισιόν γιατί για μια τέτοια κραυγαλαία περίπτωση δεν ξεκίνησε μια διαδικασία παραβίασης όταν βλέπουμε ε, τη ζημιά των τοπικών αρχών που καταγγέλουν ε, τις συμπεριφορές αυτές. Αν δεν έχετε καμία αντίρρηση, να θεωρήσουμε ότι αυτές οι τρεις πρωτοβουλίες εγκρίνονται για αυτήν την αναφορά. Ευχαριστώ τους αναφέροντες, αν δεν θέλουν κάτι να προσθέσουν και ολοκληρώνω. Θέλετε το λόγο. Θα ήθελα να πω σας ευχαριστώ, γκράτσι και ντάνκε σε όλους σας που μας πήρατε στα σοβαρά. Ευχαριστούμε. Εσάς σας ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην 1367 του 2007 που αφορά σε δύο σχέδια μεγαχωματερών σε μία γαλλική κομμόπολη. Δίνω το λόγο στην κυρία Ηλιά Νοντονή που είναι και η πρώτη υπογράφουσα. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Δεν είμαι η κυρία Οντονέ. Είμαι η Μαρή Ζωζέ Μαζίωρα, είμαι δήμαρχος ε, μιας άλλης κομμόπολης ε, που επίσης ε, πλήττεται από τη δημιουργία των δύο χωματερών. Λοιπόν, στα νότια λοιπόν των Παρισίων, ένα στεσκοπή και άλλο στον Κρολιό, η εταιρεία ΣΥΤΑ Ile de France ζήτησε την άδεια από τις κρατικές υπηρεσίες. Αν το πρόγραμμα, αν εγκαταλείφθηκε το σχέδιο των Κρολιέ, το πρόγραμμα εγκατάστασης του Σέντος Κομπίλ που θα δεχόταν απόβλητα βιομηχανικά απλά, αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας έρευνας τον Αύγουστο του 2007. Τελικά ένα έγγραφο σχεδιασμό όσον αφορά ε, τη, χωροταξία, έβαλε, την περιοχή την έβαζε σε γεωργική περιοχή και αυτή η ταξινόμηση ήταν αντίθετη με τις τοπικές κοινότητες και αποτελούσε ε, δεν επετρέπε οικοδόμηση άδεια οικοδόμησης και γι' αυτό εκπρόσωποι του, ο του κράτους θεώρησε ότι ήταν κοινοφελές το έργο κατόπιν αποφασίσεως του 13ης Μαρτίου του 2009. Οι κοινότητες ενδιαφερόμενες καθώς και η, Ένω, η εταιρεία, η Ένωση Προστασία του Περιβάλλοντος που εκπροσωπώ εξίσου αμφισβητεί το κοινοφελές αυτού του έργου βλέπει ότι δημιουργούνται πολλά προβλήματα για το περιβάλλον. Πιο γενικά λοιπόν αυτό το πρόγραμμα ε, βρίσκει αντίθετε σε όλες τις τοπικές κοινότητες ε, το Συμβούλιο της ΕΣΟΝ και το Περιφερειακό ε, Συμβούλιο της Ile de France και κινητοποιήθηκαν οι τοπικοί πληθυσμοί η επιλογή της τοποθεσίας δεν ανταποκρίνεται σε καμία ανάγκη κοινοφελούς υπηρεσίες, απλώς ε, είναι τελικά οικονομικά ωφέλη που διώκονται. Και παρόλο που δεν ενδείκνεται να εγκατασταθεί ένα κέντρο ε, αποθήκευσης αποβλήτων από την αρχή της ε, διαδικασίας, οι ντόπιοι κάτοικοι και οι κοινότητες υπογράμμισαν την ιδιαιτερότητα της τοποθεσίας, βρίσκεται στο, στον πιο σημαντικό υδροφόρο ορίζοντα όσον αφορά τον όγκο του στη Γαλλία. Και η κατάσταση υδρογεολογική δεν είναι θετική και ευνοϊκή, διότι υπάρχει κάποιο ρήγμα στην τοποθεσία και τελικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ε, μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και αυτό θα συνεπέφερε μεγάλες συνέπειες για τους, υδροφο- για τους υδατικούς, υδάτινους πόρους περιοχής. Η τοποθεσία ανήκει σε γεωργική περιοχή με εκμεταλλεύσεις ε, βιολογικών, με βιολογικές καλλιέργειες και εκεί ο κίνδυνος προβλημάτων ε, και ρήπανσης των εκμεταλλεύσεων ε, δημιουργούν βάσιμους φόβους και μπορούσαν οι ζημίες να είναι πάρα πολύ σημαντικές για τους ε, γεωργούς. Η επιλογή της τοποθεσίας δεν σέβεται καθόλου την αρχή της εγκύτητας, διότι τα απόβλητα που θα πρέπει να πάνε εκεί προέρχονται από το Παρίσι και από τα πράστια του Παρισιού, δηλαδή πάνω από 60 χιλιόμετρα απόσταση. Το ίδιο το πρόγραμμα και το έργο δεν ανταποκρίνεται σε καμία ανάγκη κοινοφελούς υπηρεσίες και για τα απόβλητα όπω είχε παρουσιαστεί. Γι' αυτό το πρόγραμμα φαίνεται αντίθετο μετά το 13 της οδηγία 2008 2008-98 ΕΟΚ που καθορίζει στόχους όσον αφορά την εξάλληψη και την κατεργασία των αποβλήτων. Τα κράτη-μέλη λέει ότι παίρνουν τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται χωρί να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρί να ενοχλείται και να επηρεάζεται αρνητικά το περιβάλλον, χωρί να δημιουργούνται κίνδυνοι για το νερό, για τον σφαιρικό αέρα, για το έδαφος, για την χλωρίδα και την πανίδα. Το πρόγραμμα αυτό για το συγκεκριμένο συγκεκριμένη τοποθεσία δημιουργεί προβλήματα και για την ατμόσφαιρα και για το έδαφος και για το νερό. Λοιπόν, η συντονισμένη δράση επέτρεψε να συλλεχθεί τεχνογνωσία και στοιχεία και ε, με επικοδομητικό τρόπο τα χρησιμοποίησαμε αυτά για να ρεβίσουμε το θέμα. Η Γαλλία δεν σέβεται τις διατάξεις της οδηγίας για τα απόβλητα του 2008 και επ' αυτού θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Γαλλία ποτέ δεν ενσωμάτωσε την οδηγία του 2008 στην ένομο τάξη της παρόλο που η προθεσμία ε, ενσωμάτωση εθνικό δίκαιο έχει εκπνεύσει. Και δείχνουν οι εμπειρογνώμονες ότι η Γαλλία ε, την 2060 δεν την εφάρμοσε για το πλαίσιο για την κοινοτική πολιτική στον τομέα των υδάτων όσον αφορά το άρθρο 4 της προαναφερθής οδηγίας, όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα, ε, τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για να αποφύγουν ή να περιορίσουν την ε, ε, απόρριψη αποβλήτων στα υπόγεια ύδατα και να αποφύγουν την επιδίνωση της κατάστασης αυτών με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 7 και την επιφύλαξη της παραγράφου 8 και την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 11 παραγράφους 3. Αυτό που αποκαλύφθηκε και ήταν εκπληκτικό ήταν η βούληση να πιέσει το κράτος να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο αποθήκης αποβλήτων και ο νομάρχης Τρεσόν ε, θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλία ε, μάλλον ανέλαβε την πρωτοβουλία κατά των κατοίκων της περιοχής και κατά των εκπροσώπων της περιφέρειας. Υπάρχει αλληλογραφία του αντιπροέδρου της περιφέρειας που έστειλε στον Ομάρχη επιστολή και, παρα... και μη εφαρμόζοντας τους νόμους που θα έπρεπε ε- έβγαλε διάταγμα νομάρχης για να καταργήσει τα εμπόδια που υπήρχαν για να δημιουργηθεί εκεί και ξεκίνησε κατηδίαν η ίδια πρωτοβουλία μια... αυτή την κίνηση για να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο εκεί παραβιάζοντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και γι' αυτό ζητούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κάθε τρόπο να παρέμβει, ούτω ώστε να, σταμα... να συμμορφωθεί με τι ευρωπαϊκέ οδηγίε το γαλλικό κράτος όσον αφορά το κέντρο αποθήκευση αποβλήτων του Σκομπί και θα θέλαμε μία αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πάει επί τόπου, ούτως ώστε να, να δει πόσο άχρηστο είναι όλο το έργο αυτό και τι συνέπειε ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει αυτό το έργο όσον αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα στην περιοχή. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Δίας Δεκαστήγιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα. Η υπόθεση αυτή ανάγεται τουλάχιστον στο 2008 Τότε έλαβε τις πρώτες πληροφορίες η Κομισιόν και έβγαλε μια ανακοίνωση. Μόλις το Φεβρουάριο φέτος έλαβα περαιτέρω πληροφορίες για την υπόθεση αυτή και ελέγχθη πως ε, θα γίνονταν δύο έργα, ένα στο Μπροσλία και ένα στο Σανσκοβίλ για ε, κατασκευή χωματερών. Με βάση τις πληροφορίες λοιπόν που λάβαμε αντιλαμβανόμαστε και διορθώστε με αν κάνω λάθος πως και οι δύο χωματερές είναι ακόμα στο στάδιο του σχεδιασμού. Οπότε η θέση της Κομισιόν τότε και τώρα είναι πως δεν έχει υπάρξει ακόμα παραβίαση της κοινωτικής νομοθεσίας. Τούτου λεχθέντος πρέπει να πούμε πως στην περίπτωση αυτή οι αναφέροντες έχουν κάνει αυτό το οποίο έπρεπε, δηλαδή ε, πήγαν στα εθνικά δικαστήρια. Όπως ξέρετε, έχουμε πολλές αναφορές. Μιλούσατε για στατιστικά πριν. Τα τελευταία τρία χρόνια εγώ έχω δει 49 αναφορές, 51 ε, γραπτές ερωτήσεις ε, και πάρα πολλές από αυτές είναι να φύγει από εδώ πέρα και ο θέλει να Οπότε Κομισιόν θα χρειαστεί δηλαδή ε, μια υπηρεσία ξεχωριστή αν είναι να ελέγξουμε κάθε περίπτωση επιτόπου. Ε, και το είπε και ο πως δεν έχουμε τους πόρους, βασιζόμαστε λοιπόν. Ε, η οδηγία δίνει την αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη να φροντίσουν να συμμορφώνονται οι χωματερέ με την κοινοτική νομοθεσία και για να είμαστε ακριβεί, μιλάμε για την οδηγία περιχητά που ανέφερε και ο συνάδελφο. Η οδηγία αυτή δεν έχει πολύ λεπτομερής διατάξεις, δηλαδή λέει πόσα μέτρα πρέπει να απέχει από οικισμούς, και αναφέρεται στην 1.2 παράρτημα 2 πως εάν ένα κράτος μέλος μετά την αξιολόγηση κινδύνου το κράτος, με συγχωρείτε, μετά την αξιολόγηση κινδύνου αποφασίζει που θα κατασκευαστεί οχητά. Όσον αφορά λοιπόν τα μέτρα μη μεταφορά τη οδηγία στο εθνικό δίκαιο από πλευρά Γαλλία. Ε, να είστε σίγουροι πως η Κομισιόν έχει σκληρή γραμμή ως προς αυτό και η προθεσμία μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 10 Δεκεμβρίου πέρσι και όσα κράτη-μέλη δεν μετέφεραν νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο <clears throat> θα διωχθούν. Θα αναλάβουμε νομική δράση από εκεί πέρα. Γι' αυτό δεσμεύομαι. Τέλος, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, η χωματερή του Γκροσλίε σταμάτησε, νομίζω, το έργο σταμάτησε μέσω δικαστικών μέσων και η χωματερή του Σανεσκοπή, τι διαβάζω εδώ πέρα, Κοιτάστε από αρμόδια δικαστήρια. Οπότε, αυτά είναι καλά νέα. Προσφύγατε στα διοικητικά δικαστήρια. Ε, Ζητήσατε λοιπόν εθνικά ένδικα μέσα Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ. Ζητάει κάποιος το λόγο. Γιάρα, ο κύριος Γιάρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ την Κομισιόν και τους αναφέροντες. Νομίζω σε ερχόμαστε σε ένα πρόβλημα αρχής που είχαμε στην Επιτροπή μας. Σωστό είναι να λέει η Κομισιόν πως υπάρχει ευρωπαϊκό δίκαιο και η εφαρμογή απευθύνεται στα κράτη-μέλη και δικαίως πάλι η Κομισιόν λέει επί της αρχής πως υποθέτουμε πως τα μέτρα και ο σχεδιασμός ε, από πλευράς κρατών μελών ε, βασίζονται στον νόμο. Αυτή είναι μία πλευρά. Η άλλη ιστορία είναι που έχουμε αναφέροντες που είναι επιφυλακτικοί και λένε δεν σας πιστεύουμε πως έγιναν όλα τόσο σωστά και η Κομισιόν λέει είναι στον προγραμματισμό, δεν μπορούμε ακόμα να κάνουμε τίποτα. Υποθέτουμε πως το κράτος μέλος θα τηρήσει νομοθεσία. Μέχρι εδώ καλά. Αλλά έχουμε, βλέπετε, και την προηγούμενη αναφορά. Πως όταν έχουμε κάποια γεγονότα μετά, όταν γίνει η χωματερή και τότε διαπιστώσουν οι αναφέροντες πως έχει παραβιαστεί το ισχύον δίκαιο, είναι δύσκολο να αναστραφεί η κατάσταση. Γι' αυτό η παράκλησή μου και εδώ πέρα η Κομισιόν στην τελευταία παράγραφο ε, ζητάει από τους αναφέροντες ε, εάν υπάρχουν πληροφορίες ε, που δείχνουν παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας να τη στείλουν στην Κομισιόν. Ναι, βεβαίως. Αυτό εγώ το θεωρώ κάποια και το συμπέρασμά μου είναι πως θα πρέπει και από πριν ε, καμιά φορά να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί, να βλέπουμε τηρείται το, το ισχύον δίκαιο. Δηλαδή να λέει η Κομισιόν βασιζόμαστε ότι τα κράτη θα τηρήσουν ε, την νομοθεσία, ε, δεν φτάνει κάπως. Και λέτε εδώ πέρα πως εάν περιέλθουν στη γνώση των αναφερόντων ε, πράγματα τα οποία είναι παραβίαση του δικαίου, να απευθυνθούν στην Κομισιόν κτλ. Τώρα από την άλλη, για να σας πω και σας κάτι, ε, και η Κομισιόν λέει πως δεν απαγορεύεται η σκέψη και ο προγραμματισμός. Ε, οπότε, σε αυτή τη δύσκολη φάση είμαι τώρα, ότι και εσείς ε, μπορείτε να κάνετε κάτι αν υπάρξει κάτι συγκεκριμένο. Οπότε πρέπει να παρακολουθείτε τα, τα πράγματα στενά. Ε, εντάξει, το, το δίκαιο ισχύει και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα αυτά συζητήσουμε. Άλλη παρέμβαση. Θα μιλήσει άλλος. Ε, δεν ζητάει άλλο το λόγο. Πιστεύω βλέποντας την παρέμβαση του συναδέλφου Γιάρο ότι είναι αρκετά ξεκάθαρη η ανάγκη που υπάρχει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην όλη προβληματική που εξέθεσαν οι αναφέροντες. Πιο συγκεκριμένα πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον έκανε την ανάλυση μόνο ενός τμήματος του προβλήματος που εφήγει διότι είναι και θέμα παραβίασης, όχι μόνο μη ορθής εφαρμογής της οδηγίας για τα απόβλητα, για το περιβάλλον. Ε, υπάρχουν διάφορες στοιχές που πιστεύω ότι θα πρέπει να εξεταστούν σε μεγαλύτερο βάθος από ό,τι έγινε μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή μας να εξετάσει εις βάθος το γεγονός που αναφέρεται και την υπόθεση αυτή και αναμένεται γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Εκτελεστική Επιτροπή, που ακόμα δεν κατέφθασε. Η απάντηση που εδόθηκε εδώ θα πρέπει να ακολουθηθεί με πληρέστερο τρόπο να δοθούν και άλλα στοιχεία που ελήφθησαν και παρελήφθησαν πιο πρόσφατα, όπως είπε εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δοθεί κάποια κοινοποίηση και στι εθνικές εθνικέ αρχέ, ώστε μαζί με τι εθνικέ αρχέ να γίνει μια αξιολόγηση, να, γνωστοποιηθεί ότι ε, ίσως θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες που γίνονται σε, αυτή την, ε, σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις, εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις και αν δεν υπάρχει λόγος θέλετε να ε, δευτερολογήσετε, συγγνώμη από την κυρία Δήμαρχο, που δεν σας ανέφερα σωστά, σας σύστησα σωστά. Θέλετε κυρία Δήμαρχε να πείτε κάτι. Ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών που εξέτασε την υπόθεσή μας και ελπίζω ότι αυτό θα βοηθήσει ενδεχομένως και άλλες ενώσεις και άλλους που έχουν προβλήματα με τέτοιες χωματερές, ούτως ώστε να εμποδιστεί η ύπαρξή τους και η δημιουργία τους πριν μολύνουν. Είναι πολύ σημαντικό ε, και θέσατε σωστά και θίξατε σωστά το πρόβλημα και σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ εσάς. Πάμε στο επόμενο σημείο, την Επιτροπό 13-18-2008 που αφορά μη συμμόρφωση προς την ομεθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το περιβάλλον σε σχέση με την εξόριξη αδρανών υλικών κοντά σε περιοχή του δικτύου Natura 2000 στη Νότια Πολωνία. Δεν είναι παρόν ε, εκείνος που υπέγραψε την αναφορά, οπότε θα δώσω αμέσως το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τσιπριάνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην αναφορά αυτή ήδη έχουμε βγάλει τρεις ανακοινώσεις, τελευταία ήταν το Σεπτέμβριο του 2010. Αναφέρον, παραπονιόταν για ζημιές που προκαλούσε στο περιβάλλον η εξόριξη αδρανών υλικών σε ένα λατομείο, σε ένα σημείο που είχε καθοριστεί ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με την οδηγία βιοτόπων. Αξιολογήσαμε λοιπόν την κατάσταση υπό το φως διαφόρων διατάξεων της οδηγίας περί η άδεια εξόριξης δόθηκε το 1999, πολύ πριν την ένταξη της Πολωνίας και πολύ πριν οριστεί το συγκεκριμένο μέρος ε, ε, ως τοποθεσία σημασία σύμφωνα με την οδηγία βιοτόπων. Αυτό έγινε το 2008. Άρα η διαδικασία και κανόνες σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας δεν ίσχυαν όταν δόθηκε άδεια. Αυτό το οποίο ίσχυε όμως ήταν οι διατάξεις του άρθρου 6 παραγραφός 2 της οδηγίας που λέει πως τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν, να κάνουν ενέργειες για την ε, μη ε, επιδίνωση του βιοτόπου των ειδών και εκεί πέρα καλύπτονταν και η συγκεκριμένη τοποθεσία. Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες που μας έδωσαν οι πολωνικές αρχές, συμπεραίνουμε πως οι πολωνικές αρχές έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να αναστείλουν την άδεια εξόριξης άδρανων υλικών. Ενημερωθήκαμε μάλιστα από την Πολωνία πως οι εξορυκτικές δραστηριότητες σταμάτησαν το 2009. Οπότε το θέμα παραβίασης ε, του άρθρου 6 παραγραφος 2 της οδηγίας περί ποιοτόπων έχει ήδη αντιμετωπιστεί. Όσον αφορά την ε, πιθανή μελλοντική επέκταση της, ε, του λατομπίου, αυτό δεν, δεν έχουν δώσει σχετική άδεια ακόμα οι αρχές και εάν οι πολωνικές αρχές θέλουν να δώσουν τέτοια άδεια, οι κανόνες και οι διαδικασίες της σχετική οδηγίας, δηλαδή το άρθρο 6 παράγραφος 2 εδώ πέρα, και τι οδηγίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ο συνάδελφο Βίλαντ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Έχει μπλοκαριστεί το σχέδιο και έχουν περιοριστεί και οι ζημιές στο περιβάλλον. Τώρα θα πρέπει να επέμβουμε για να επανορθώσουμε την κατάσταση. Και όσο δεν συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά το θέμα. Νομίζω ότι είναι σαφέστατα τα πράγματα. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Βαλέσσα. Συγγνώμη, συγγνώμη που έκανα λάθος το όνομά σου. Θέλει κανείς άλλο το λόγο, όχι. Παραμένει ανοιχτή η αναφορά. Είναι ανοιχτό το θέμα και για την Κομισιόν. Η Κομισιόν μας ανέφερε ότι έχουμε έναν διάλογο μερικός παραγωγικό με τις πολωνικές αρχές. Θα περιμένουμε λοιπόν. Επόμενη αναφορά 944-2009 που αφορά στο έργο εξόριξης πετρελαίου στον προστατευόμενο δρυμό της ε, Βάλεντελ κουρώνε Δίνω το λόγο στον δόκτορα Τσίπριάνη σχετικά. Ευχαριστώ ότι αυτή η περιπτώση ο αναφέρον διαμαρτυρόταν για το πρόγραμμα για μια εγκατάσταση για γεώτρηση για πετρέλαιο που υποτίθεται θα πήγαινε στο πάρκο Μοντεβέκιο στο πάρκο του Παλώνε που ήταν σημαντικός τόπος στα πλαίσια της οδηγίας για τους βιοτόπους Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν απάντησε στον αναφέροντα είπε ότι εν τη αυτή περιπτώση η οδηγία περί και σχετικές διαδικασίες που αφορούν την, την οδηγία για την αξιολόγηση συνεπιών ήταν διατάξεις που ίσχυαν αλλά δεν μπορούσε να εντοπιστεί παραβία στον λόγο διατάξεων διότι είχε δοθεί, δεν είχε δοθεί ακόμα άδεια για κάτι τέτοιο. Έκτοτε δεν παραλάβαμε άλλες πληροφορίες από τους αναφέροντες για το έργο, αν εξετελέστη ή όχι, αν ενεκρίθη ή όχι. Δεν λάβαμε καμία άλλη διαμαρτυρία, καταγγελία για την υπόθεση αυτή. Ερευνήσαμε και επίσης στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες για να βρούμε άρθρα. Ανεπίσημα ήρθαμε σε επαφή με τις περιφερειακές αρχές και ανακαλύψαμε ότι αυτό το έργο απεσύρθη από την πετρελαϊκή εταιρεία, η πρόταση αυτή είδε τον Αύγουστο του 2009. Ένα μήνα μετά την υποβολή της αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά από μαζική κινητοποίηση των ντόπιων που διαμαρτυρόταν για αυτό το πρόγραμμα, για αυτό το έργο. Γι' αυτό το πρόγραμμα αυτό εγκατελείφθη και δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε κάποια παραβίαση της νομοθεσίας της σχετικής για το περιβάλλον. Υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις, θέλει κάποιος να πει κάτι. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Βάσει λοιπόν αυτή τη ανακοινώσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, η πρότασή μου θα ήταν να κλείσουμε την αναφορά αυτή με μόνη επιφύλαξη μία επαλήθευση ίσως και άτυποι με το αναφέροντα μέσω της γραμματείας. Μέσω ε, με μία ανταλλαγή απόψεων να εξακριβωθούν αν είναι σωστά τα στοιχεία που δόθηκαν και αν ισχύουν αυτά που να την αναφορά. Πάμε λοιπόν στην αναφορά 12, του σημείου 12, 1833 του 2008 που αφορά μία πιθανή κρατική ενίσχυση στην, ε, στην Κασάνδρα και την πώληση των μεταλλίων Κασάνδρας στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Δίνω το λόγο στον Δημήτριο Πύλιο που είναι και ο υπεύθυνο εκ μέρους της Κομισιόν. Ότιμη κυρία Πρόεδρε, ε, στις 23 Φεβρουαρίου του 2011 ύστερα από μια επίσημη διαδικασία έρευνας η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2008, η Επιτροπή έφτασε στο... Παρακαλώ. Η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφτασε στο συμπέρασμα ότι η πώληση των μεταλλίων Κασάνδρας από το ελληνικό δημόσιο προς την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, η οποία έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2003, έγινε σε τιμή χαμηλότερη από την αγοραία αξία των ε, μεταλλίων. Η πώληση αυτή είχε γίνει χωρίς τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ή την εκτίμηση της αγοράς αξίας των ε, πολυθέντων περιουσιακών στοιχείων από ανεξάρτητο εκτιμητή. βασιζόμενοι σε εκτίμηση της αγοράς αξίας των, περιουσιακών, ε, των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, η οποία έγινε αμέσως μετά την πώληση ε, για λογαριασμό της ε, εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, η Επιτροπή τοποθέτησε την αγοραία αξία των ε, πολυθέντων μεταλλίων στα 25 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σε 14 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από την τιμή στην οποία απολύθηκαν. Ταυτόχρονα το, η Σύμβαση Πώλησης προέβλεπε την απαλλαγή από φόρους επί της συναλλαγής ύψους 1,34 εκατομμυρίων ευρώ Επίσης, η Επιτροπή έφτασε στο συμπέρασμα ότι τα συγκεκριμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων δεν ήταν συμβατά με την συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, έφτασε η Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός εποφελήθηκε από μη συμβατές κρατικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 15,34 εκατομμύριων ευρώ, τις οποίες θα πρέπει η Ελλάδα να ανακτήσει με τους προβλεπόμενους τόκους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Αλαβράκα. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τις απόψεις της Επιτροπής και διάβασα όμως εν τω μεταξύ την από 20 του 2000 αναφορά της Επιτροπής ε, προς ε, ε, την δική μας Επιτροπή. Βλέπω ότι στο ιστορικό αναφέρεται ότι αγόρασε στις 12 Δεκεμβρίου του 2003 το ελληνικό δημόσιο αντί ποσού 11 εκατομμυρίων ευρώ το όλον συγκρότημα των μεταλλίων Κασάνδρας και το πούλησε την ίδια ημέρα αντί του ιδίου τιμήματος των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό με προβληματίζει νομικά. Πρώτον, εάν και κατά πόσον ή το δυνατόν να γίνει μεταβίβαση την, την ίδια μέρα διότι υπάρχουν ε, θέματα κυριότητος τα οποία πρέπει να μεταγραφούν και δεν προλαβαίνει σε μία μέρα να γίνει μεταγραφή και η πώληση, πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Και δεύτερον διότι τα 11 εκατομμύρια ευρώ τα πήρε το ελληνικό δημόσιο, τα κατέβαλε όπως το λέει η έκθεση της Επιτροπής, τα κατέβαλε και τα πήρε την ίδια μέρα. Άρα δεν κατέβαλε. Πήρε τα ίδια χρήματα. Δεν κατανοώ λοιπόν γιατί να πρέπει να κερδοσκοπεί το ελληνικό δημόσιο ή οποιοδήποτε δημόσιο εις βάρος της προκτήτωρος TVX. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ότι υποθάλπεται μια κακή κερδοσκοπία του ελληνικού δημοσίου ή οποιοδήποτε δημοσίου κατά μια εταιρεία που έχει πτωχεύσει. Άρα ή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η εταιρεία TVX, η ιδιωτική εταιρεία, η οποία εστερήθη των περιουσιακών στοιχείων και στην ουσία το τίμημα το έλαβε από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός την ίδια μέρα με την παρεμβολή αυτή του ελληνικού δημοσίου, την περίεργη, δεν ξέρω πώς είναι, και γι' αυτό θα ήθελα χρόνο να το εξετάσουμε, ή θα πρέπει να πούμε ότι υποθάλπουμε κερδοσκοπίες των δημοσίων εις βάρος ιδιωτών. Υπό τα δεδομένα αυτά θεωρώ ότι δεν μπορώ να αποφασίσω για να δω και να εκφράσω άποψη ή αν κατά πόσο ευσταθεί η και κατά πόσον ευσταθεί η άποψη αυτή της Επιτροπής και θα ζητούσα χρόνο να το εξετάσουμε και εμείς και εσείς και να δούμε και το γενικότερο θέμα της κερδοσκοπίας των κρατών εις βάρος ιδιωτικών εταιριών οι οποίες πτωχεύουν ή τις οδηγούν σε μια πτώχευση. Πολύ περισσότερο όταν σε, ένα κράτος όπως είναι η Ελλάς και, όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητάνε επενδύσεις αυτή τη στιγμή. Σημειώνω ότι έχω ιδιαίτερες αντιθέσεις σαν ε, πολιτικός και σαν ε, πολιτικό σχήμα εναντίον της γίνει ιδιοκτήτριας των ε, μεταλλίων της Κασάνδρας αλλά αυτό δεν, δεν μου επιτρέπει να μεροληπτήσω εις βάρος της. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να το δούμε το θέμα, να κρατηθεί ανοιχτή και να ζητηθούν αυτά ακριβώς τα στοιχεία εκ μέρους των ελληνικών αρχών αλλά και της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ναι. Ε, ναι, ε, από την ημερομηνία που ε, έβγαλε η Επιτροπή η Κομισιόν την απόφασή της, είχατε καμία αντίδραση από το ελληνικό δημόσιο, από, την ελληνική πολιτεία. υποθέτω ότι μπορώ να σας πω πως όχι. C'era prima la collega Zanoca. Η Kiria Γερόκα. But I just wanted to ask the... Θέλω να ρωτήσω ε, επί της διαδικασίας και το σύνολο των ε, αναφορών που έχουμε τώρα. Που έχουμε έξι αναφορές Δεν ξέρω αν έχουν κάτι να πούν οι συνάδελφοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα περιμένω εγώ. Γιατί μία, μία ερώτηση έχω και κατά βάση είναι αντίρρηση της διαδικασίας για όλες αυτές τις ε, αναφορές που ερευνήσαμε. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πιο αιτιολογημένες απαντήσεις από την Κομισιόν. Όλες οι απαντήσεις που έχουμε εδώ πέρα είναι παλαιότερες. Και τώρα έχουμε κάποιες δηλώσεις με νέες πληροφορίες από την Κομισιόν που στην προηγούμενη παραδείγματος χάρη αναφορά αλλάζει τελείως την κατάσταση. Δεν ξέρω. Είμαστε στο Μάρτιο του 2011 και έχουμε απαντήσει εδώ πέρα του 2008-2009 πιο πρόσφατη είναι του 2010. Είναι δυνατόν να έχουμε πιο πρόσφατες αξιολογήσεις κατάστασης. Αλλιώς ε, εξετάζουμε περιπτώσεις οι οποίες είναι ε, δηλαδή, στις οποίες η κατάσταση έχει αλλάξει και δεν έχει νόημα να τη συζητάμε. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε από την απάντηση που η Κομισιόν έδωσε στην κυρία Παλιαδέλη αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει υπόψη της αντίδραση του ελληνικού δημοσίου. Είναι ορθό. Όμως παρά τα αυτά εγώ γνωρίζω ότι η απάντηση της από 24 Δευτέρου 2011 απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκδόθηκε στις 11 Τρίτου του 2011 από το αντίστοιχο Υπουργείο αντιρρητική, αντιρρητικό έγγραφο στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ το ελληνικό δημόσιο αμφιβάλλει τόσο για την ακρίβεια όσο και για την ουσία των επιχειρημάτων της ε, Επιτροπής. Επομένως, ε, έγγραφο το οποίο μπορώ να θέσω υπόψη σας, αν δεν έχετε άλλο τρόπο να το αποκτήσετε. Επομένως, κυρία Πρόεδρε, θα συμφωνούσα με τον κύριο Σαλαβράκο ότι θα έπρεπε να γίνει μια ε, συζήτηση γιατί μου φαίνεται ότι εδώ, χωρίς να είμαι δικηγόρος, υπάρχει μια διχογνωμία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές αρχές και στην ερμηνεία που αποδίδουν σε διάφορες νομικές πράξεις και του ελληνικού δημοσίου που αντιτίθεται και λέει ότι η Επιτροπή δεν τα εφαρμόζει, δεν τα κατανοεί καλά. Θα μπορούσα να σας διαβάσω εδώ ένα σημείο μόνο ε, στο οποίο λέει το ελληνικό δημόσιο αποφαίνεται ότι η μελέτη η οποία υπέβαλε στην Επιτροπή ο καταγγέλων της πώληση από την εταιρεία Μπέλε και Ντόλμπερ, η ελληνική πολιτεία ισχυρίζεται πως είναι λανθασμένη και πως δημιουργεί εντυπώσεις για τους παρακάτω λόγους και εκθέτει τους λόγους. Σε άλλο σημείο εκθέτει άλλο πράγμα. Επομένως νομίζω ότι αυτή η υπόθεση, για να μην μακρηγορώ, μια που δεν είμαι και νομικός κιόλα, θα άξιζε τον κόπο περαιτέρω να συζητηθεί επί των πραγματικών δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ συνάδελφοι. Νομίζω ότι είναι αρκετά ομόφωνο το αίτημα να εμβαθύνουμε περαιτέρω και να έχουμε και μία γραπτή ανακοίνωση με περισσότερα επιχειρήματα και πιο διαρθρωμένη εκ μέρους της Κομισιόν από αυτή που ακούσαμε σήμερα, διότι έχουμε αντιρρήσεις και τεκμηριωμένες αντιρρήσεις. Και θεωρεί η Κομισιόν ότι η Επιτροπή μας, συγγνώμη, θεωρεί ότι υπάρχουν λόγοι να θεωρείτε ότι συνεχίζεται η παραβίαση, οπότε θα πρέπει να συνεχίσει και η Κομισιόν τη δική της διερεύνηση. Συμφωνούμε. Κλείνουμε τη συζήτηση για αυτή την αναφορά. Η συνάδελφος Παλιαδέλη. τουλάχιστον και η Επιτροπή ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εγγράφου του ελληνικού δημοσίου για το οποίο μας μίλησε ο κύριος ε, Τσουκαλάς λίγο πριν λίγο. Επομένως, ε, εφόσον έτσι επιθυμείτε, προφανώς έτσι θα γίνει. Ωραία, ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν. Στην επόμενη αναφορά, 931 ε, κάθετος 2009, σχετικά με την εικαζόμενη κατάχρηση χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, έργο, για ένα έργο υποδομής στην πόλη του Νικηφόρου. Είναι παρόν ο υπογράφων, είναι ο Νικόλος Καγιαογλού, ο οποίος είναι και ο δήμαρχος του Νικηφόρου και συγγνώμη για το πώς ε, πρόφερα το όνομά σας. Καλησπέρα στην Επιτροπή. Ε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε αυτό το αίτημα να το φέρουμε εδώ και να το συζητήσουμε. Ονομάζομαι Σπύρος Λάτσας, είμαι δημοσιογράφος και εκπροσωπώ εδώ δίπλα μου τον ε, δήμαρχο του Δήμου Παρανεστίου, του πρώην Δήμου Νικηφόρου, τον κύριο Νίκο Καγιάογλου. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι έχουμε προσφύγει στην Επιτροπή σας γιατί έχουμε διαπιστώσει, έχει διαπιστώσει ο Δήμαρχος και ο σημερινός Δήμαρχος, τότε Δημοτικός Σύμβουλος, σε ένα έργο το οποίο εκτελέστηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να είμαι πιο σαφής με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην όμως εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν και γεγονότα τα οποία συνέβησαν εκεί δεν ε, τηρήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Ουσιαστικά δηλαδή με δύο λόγια θα σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε μία συγχρηματοδότηση 75% σε ένα ύψος ποσού 300.000 ευρώ πλην όμως αυτό δεν ε, έγινε σύμφωνα με την προβλεπόμενη μελέτη. Ο κ. Καγιάγλου τότε ως ε, δημοτικό Σύμβουλος ε, απευθύνθηκε σε πάρα πολλές ε, ελληνικές αρχές. Δυστυχώς όμως δεν ξέρω τον τρόπο και για ποιο λόγο έγινε αυτό. Οι πόρτες δεν ήταν και πάρα πολύ ανοιχτές δεδομένου ότι στη χώρα μας και λυπάμαι που το λέω αυτό, σε πολλές των περιπτώσεων υπάρχει μια αλληλοκάλυψη αν θέλετε των υπηρεσιών και δι' όταν πρόκειται για τεχνικές υπηρεσίες. Θέλω λοιπόν να σας πω και αναφερόμενος πάντα στην ε, αναφορά στην 931 ε, αυτή που συζητάμε ότι για το συγκεκριμένο έργο έχουν ε, βεβαιωθεί τεράστιες αποκλήσεις από την αρχική εγκεκριμένη μελέτη, περιβαλλοντικές βλάβες σημαντικές, παράβαση ουσιοδών διατάξεων νόμων περί κολλημάτου συμφέροντος και θα σας εξηγήσω γιατί, καθώς όπως σας είπα και εργασίες που πληρώθηκαν χωρίς να έχουν εκτελεστεί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή εδώ η αναφορά η οποία γίνεται έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι τα χρήματα τα οποία διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χώρα μα ε, για να εκτελεστεί ένα έργο το οποίο είναι έργο ίδρυυση και μάλιστα ο τίτλο του είναι Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυση στη θέση νικηφόρου, του πρώην Δήμου Νικηφόρου, ε, στη θέση πηγών Βάγια. Και το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με το ηθικό ασυμβίβαστο, αν θέλετε, ή με το κόλλημα συμφέροντο είναι ότι ο προϊστάμενος τη εν λόγω υπηρεσία, τη τεχνική υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων είναι συγγενής, πρώτου βαθμού, συγγενής μάλλον, με την ε, κυρία η οποία έχει αναλάβει το έργο. Δηλαδή πρόκειται για μια οικογένεια η οποία έχει ε, καθόλου ανώμημα βέβαια, καθόλου ανώμημες έχουν τηρηθεί οι διαδικασίε, τουλάχιστον ή αν θέλετε νομιμοφανεί. Έχουν λοιπόν τηρηθεί όλα αυτά και ο κύριο ο οποίο υπογράφει τα εντάλματα είναι κουνιάδος της κυρίας η οποία εκτελεί. Και θέλω εγώ να ρωτήσω την κοινή λογική, την απλή, έτσι, την, απλή κοινή λογική, εάν είναι δυνατόν ε, ένας ο οποίος έχει το συγγενή του και εκτελεί ένα έργο, εάν είναι δυνατόν να είναι απόλυτα αμερόληπτος, εάν είναι δυνατόν να μπορεί να τηρήσει τη διαδικασία και το λέω αυτό γιατί έχει διαπιστωθεί μέσα από μία σειρά εγγράφων ότι δεν έχουν τηρηθεί όλα αυτά και θα γίνω και πιο σαφής όσο μπορώ σύντομα γιατί ο χρόνος που μου δίνεται είναι μόνο πέντε λεπτά. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής ότι ο κ. Καγιάγλου απευθύνθηκε στον ΕΣΠΕΛ, στον Ειδικό Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου, ο οποίος ε, έχει σύμβαση, είναι ισπανική εταιρεία και έχει σύμβαση με, την, με Έλληνες ε, μηχανικούς. Ο ΕΣΠΕΛ λοιπόν ήρθε και κατέγραψε μία σειρά από γεγονότα εκεί που είδε και κατέταξε το έργο στην κατηγορία 2. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένα έργο κατατάσσεται στην κατηγορία 2 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και με την κοινή υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί για τον ΕΣΠΕΛ ε, δεν μπορεί να γίνει οριστική παραλαβή του έργου. Έγινε οριστική παραλαβή του έργου διότι απεκρύπτει από το, ε, από το Δημοτικό Συμβούλιο η όχληση η οποία προσεκόμισε η, ανα, η ανάδοχος, η κυρία η οποία έκανε το έργο. Δεν έγινε αυτό η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την νομοθεσία πάλι και την κοινή υπουργική απόφαση, λέει ότι όταν όταν ένα έργο ε, έχει παρέμβει ο ΕΣΠΕΛ και το έχει κατατάξει στην κατηγορία 2 και 3 πρέπει να στείλει τις τεχνικές αναφορές στο αρμόδιο Υπουργείο, πράγμα το οποίο δεν έγινε, ούτε αυτό έγινε και όλα αυτά και άλλα πολλά που μπορώ να σας πω αν είχα παραπάνω χρόνο, ε, γιατί θέλω να καταλήξω κάπου. Όλα αυτά λοιπόν συντελούν στο ότι πραγματικά δεν μπορεί να γίνει απερίσπαστη, ή ε, αμερόληπτη αν θέλετε διαδικασία όταν ο κουνιάδος υπογράφει ε, στην κουνιάδα, να το πω έτσι απλά. Ο συγγενής στη συγγενή. Να σας πω επιπροσθέτως ότι όταν έγινε η δημοπρασία του έργου, καθόλου ανώμημη, καθόλου ε, ήταν τρεις οι, αναθε... τρεις οι εταιρείες οι οποίες ε, δώσανε διαγωνισμό, διαγωνιστική διαδικασία. Η μία εταιρεία, αυτή που πήρε το έργο, με ποσοστό έκπτωση 2,16% είναι η κυρία Βακαρτζή, η οποία πραγματικά μέσα από νόμιμες διαδικασίες πήρε το έργο. Η δεύτερη εταιρεία ήταν η εταιρεία Δία Σεβετέ, η οποία δεν είναι κουνιάδα του του προϊσταμένου της Εθνικής Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων είναι η γυναίκα του. Και η τρίτη εταιρεία, επιτρέψτε μου και ζητώ συγγνώμη για το χαρακτηρισμό, ήταν ο λαγός της υπόθεσης, ο οποίος μπήκε μέσα με 1% προκειμένου να φύγει για να μείνουν οι άλλες δύο και κάποια από τις δύο να το πάρει. Δηλαδή καθαρά οικογενειακή υπόθεση. Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο, γιατί περνάει ο χρόνος και θέλω να σεβαστώ απόλυτα όλα αυτά τα οποία είπα, ε, έτσι είπαμε από την αρχή. Θέλω μόνο να σας πω το εξής. Ζητάμε από την Επιτροπή ο κ. Καγιάγλου, Δήμαρχος Παρανεστίου, την παρέμβασή της προκειμένου να βρεθεί μια λύση, να εκτελεστεί το έργο, διότι το έργο εκτός του ότι δεν εκτελέστηκε καθόλου και σύμφωνα με αυτά τα οποία ε, αναφέρει η τεχνική προδιαγραφή, έχει περάσει, έχει κατασκευαστεί ουσιαστικά μέσα σε χήμαρο, έχουν γίνει τρομερές περιβαλλοντικές καταστροφές, έχει παρέμβει το δασαρχείο της Καβάλας και έχει επιβάλει, αν θέλετε, έχει κάνει εισήγηση προς την εισαγγελία για μια χρηματική αποσημείωση 6.500 ευρώ για την παράνομη υλοτόμηση και 2.000 ευρώ για την ηθική βλάβη και από εκεί και πέρα κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή κάποια χωριά να μείνουν, κάποιες περιοχές να μείνουν χωρίς νερό διότι πολύ απλά θα σας πω μόνο ένα τεχνικό στοιχείο της μελέτης. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει και γι' αυτό κοστίζει 300 χιλιάρικα ότι αυτά τα 4.350 μέτρα έπρεπε να γίνουν με τα χέρια ε, με χειρονακτικό τρόπο. Γι' αυτό και ήταν τόσο πολλά τα χρήματα. Για να γίνει αυτό έπρεπε να σκαφτεί τάφρος 1,5 μέτρο επί 50 εκατοστά, να μπει άμμος από κάτω, να μπει σωλήνα από πάνω και από πάνω να εγκυβωτιστεί με τσιμέντο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δεν γίνανε και αυτό που σας λέω ε, θα σας το δώσω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας πλήρης φάκελος εδώ, ο οποίος θα κατατεθεί από τον κύριο Καγιάγλου στην Επιτροπή σας ε, και θα δείτε ότι πραγματικά η σωλήνα σε πολλές περιπτώσεις είναι 10 πόντους, σε άλλες είναι 20, σε άλλες είναι 30 και φυσικά είναι στο χώμα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν και ο πιο αδαής περί των τεχνικών ζητημάτων ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει εφαρμοστεί η τεχνική μελέτη όπως το από την αρχή και να σας πω βέβαια ότι πάρα πολλοί κάτοικοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς νερό έχοντας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσείς δηλαδή, εδώ, εμείς όλοι, γιατί μια οικογένεια είμαστε, θέλω να το πω έτσι, έχοντας δώσει λοιπόν κάποια χρήματα και έχοντας συγχρηματοδοτήσει ένα έργο. Αυτά ήθελα να σας πω. Ε, θα σας υποβληθεί πλήρης φάκελος ε, με όλα τα τεχνικά στοιχεία και θα σας πω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικηφόρου σε χθεσινή του συνεδρίαση ε, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην παραλάβει το έργο, οριστική παραλαβή και αποφάσισε επίσης να κάνει και ανάκληση του ανακεφαλαιτικού πίνακα πίνακα, ο οποίος ανακεφαλαιωτικός πίνακας, μπαίνω σε λίγο σε μια τεχνική λεπτομέρεια, έχει να κάνει σαν ένα προτιμολόγιο εργασιών και χρημάτων, έχει αλλάξει βέβαια κατά πολύ οι επιβλέποντε έχουν αλλάξει αυτόν τον χρηματοδοτικό κατάλογο, έχουν αλλάξει ως προς τι εργασίε, δεν τον έχουν αλλάξει όμως ως προς τα χρήματα. Με αποτέλεσμα, ενώ το έργο ήταν 4.350 μέτρα να γίνει με χειρονακτικό τρόπο, έχοντας 200.000 από αυτά τα χρήματα σε ημερομίσθια, Εντούτοι δεν έγινε, έγινε με μηχανικό τρόπο, κατεστράφει το δάσο, κατεστράφει το περιβάλλον, ε, δεν ξέρω αν είναι περιοχή Νατούρα δεν το έχω προλάβει να το δω γιατί είμαι συνεχώς στα δικαστήρια επειδή έκανα μια αναφορά στην εφημερίδα μου και τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να αποδείξω ότι αν και έχω κάποια κιλά δεν είμαι ελέφαντας εν πάση περιπτώσει να κάνουμε και λίγο χιούμορ και να σας πω λοιπόν ότι μόλις διαπιστώσω ότι είναι Νατούρα θα, γιατί μάλλον πρέπει να είναι Νατούρα θα ενημερώσω την Επιτροπή σας προκειμένου να καταλήξετε σε ένα πιο ασφαλέ συμπέρασμα Κλείνοντα. θέλω να σας παρακαλέσω όχι να κυνηγήσετε τον άνθρωπο αυτόν. Ε, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα κατά κόρον. Ε, οι τεχνικές υπηρεσίες των ε, Δήμων, των Ομαρχιών και εν πάση περιπτώσει όλοι αυτοί που εμπλέκονται στα δημόσια έργα είναι πολύ, πολύ λίγο γνωστό τι γίνεται. Εμείς θέλουμε να γίνει το έργο, θέλουμε τη δική σας παρέμβαση προκειμένου να αποκατασταθεί το περιβάλλον και θέλουμε εν πάση περιπτώσει να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να λειτουργούν κατά το δοκούν με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και αν έχουν ασυμβίβαστο, που έχουν δικαίωμα βέβαια και αυτοί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι και οι οικογένειές τους να δουλεύουν, και να ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα να βρεθούν δικλείδες ασφαλείας τέτοιε, οι οποίε βέβαια δεν αφορούν την Επιτροπή σα, αφορούν το εθνικό δίκαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει μια εισήγηση μπορεί να γίνει από εσά, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε ένα θέμα ότι δεν πρέπει να γίνεται κατα... κατασπατάληση του δημοσίου ευρωπαϊκού και, ελληνικού χρήματο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστούμε και εμεί. Ναι. Ναι. Επιτροπή δεν είπατε. Τότε για την, για την Επιτροπή ο κύριος Περουλάκης. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. έχει ερευνήσει το θέμα. Βέβαια, με βάση την αρχή της επικουρικότητας, η υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι οποίες κυρίως χρηματοδοτούνται μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία, βασίζεται σε μια εταιρική σχέση μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Η Επιτροπή εγκρίνει μεν τα μεγάλα έργα, αλλά όχι όμω μικρότερα έργα τα οποία είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο το οποίο καθορίζουν οι σχετικοί κανονισμοί. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι σχετικά με του ελέγχου οι προσπάθειε πρέπει να επιμερίζονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών, του κράτου μέλου και τη Επιτροπή, έχοντα κατά νου ότι η προσπάθεια πρέπει να ανάλογη και με τι δημοσιονομικέ του επιπτώσει. Βέβαια, όπου υπάρχει υποψία απάτη, εκεί η αρχή μα είναι μηδενική ανοχή. Με βάση την καταγγελία την οποία λάβαμε, ζήσαμε πληροφορίε από τι αρμόδιε εθνικέ αρχέ, και λάβαμε απαντήσεις οι οποίες περικλείουν επίσης και τον, ε, την έκθεση ελέγχου στην οποία προέβη ο ΕΣΠΕΛ. Ο ΕΣΠΕΛ είναι εξειδικευμένο σύμβουλο ποιοτικών ελέγχων, συμβουλευτικό οργανισμό που ορίστηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών μετά από ανοιχτό διαγωνισμό και έχει σκοπό να ελέγχει την ποιότητα τη εκτέλεση των δημόσιων έργων στην Ελλάδα. Ο ΕΣΠΕΛ λοιπόν κατέληξε σε μια σειρά από συμπεράσματα τα οποία κυρίω ε, επιβεβαιώνουν μια σειρά από αστοχίε σε σχέση με την τεχνική εκτέλεση του έργου, η οποία δεν, δεν ήταν ε, συναφής με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Ε, σε σχέση με το θέμα ε, της πιθανής εμπλοκής συγγενών και μιας διαδικασίας η οποία δεν θα ήταν νόμιμη ο ΕΣΠΕΛ κατέληξε ότι δεν υπήρχε τουλάχιστον στις διαδικασίες επιλογής των εργολάβων συγγενής εργολάβου ε, ε, στην Επιτροπή η οποία ενέκρινε και τη σύμβαση του έργου. Βέβαια από εκεί και πέρα ήρθε μια σειρά από δειγματοληπτικούς ελέγχους οι οποίοι επαλήθευσαν ότι όντως υπήρχαν παραβιάσεις σε σχέση με το αρχικό φάκελο και με τις αρχικές προδιαγραφές του έργου στην τελική εκτέλεση και ως εκ τούτου ο ΕΣΠΕΛ προέβησε μια σειρά από συστάσεις τις οποίες όφιλε η αρμόδια αρχή να εκτελέσει, να ειδοποιήσει τον ΕΣΠΕΛ ότι τις εκτέλεσε και μετά ο ΕΣΠΕΛ θα εξέδιδε μια καινούρια έκθεση η οποία θα μπορούσε να μας δώσει τη δυνατότητα να προβούμε στην τελική πληρωμή του έργου γιατί το έργο ε, ανήκε στην, στο <clears throat> επιχειρησιακό πρόγραμμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την περίοδο 2006 για το οποίο έχουμε ήδη λάβει την τελική έκθεση και το έργο αυτό έχει καταταγεί στην κατηγορία των ημιτελών έργων, το οποίο σημαίνει ότι δεν πληρώνουμε εξ ολοκλήρου τη συμμετοχή μα. Πληροφοριακά σα αναφέρω ότι έχουμε πληρώσει από 307.000 προπολογισμό το έργο, η κοινωνική συνδρομή που έχει πληρωθεί μέχρι στιγμή είναι 180.000, 087 ευρώ. <clears throat> Η θέση μα είναι ότι αυτή τη στιγμή το έργο είναι ημιτελές, το έργο οφείλει να αποκατασταθεί με εθνικού πόρου πλέον και από εδώ και μπρος θα πρέπει να γίνει με βάση τις ε, υποδείξεις του ΕΣΠΕΛ. Αν γίνει χωρίς ε, να σεβαστεί τις υποδείξεις του ΕΣΠΕΛ θα παραμείνει ως έχει και ως εκ τούτου θα είναι υποχρεωμένοι υποχρεωμένες οι εθνικές αρχές να επιστρέψουν το σύνολο της κοινωνικής συνδρομής που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα. Η προθεσμία για, την, ε, για τις εθνικές αρχές να υποβάλουν τελική έκθεση υλοποίησης του έργου είναι η 31 του 2012. Μέχρι τότε εμείς δεν μπορούμε να ξαναπαρεύουμε. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι στα χέρια των εθνικών αρχών. Όντως όπως ανέφερε ο καταγγέλων υπάρχει μια ε, παραλαβή οριστική του έργου η οποία δεν είναι συμβατή με τους ισχύοντες κανόνες αλλά παρόλα αυτά το έργο παραμένει στην κατηγορία 2 έχει καταταγεί στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με το οποίο παρακολουθούν οι εθνικές αρχές και η Επιτροπή την εκτέλεση των έργων παραμένει στην κατηγορία 2, δεν μπορεί να αποπληρωθεί το έργο και δεν θα αποπληρωθεί εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση με τις ε, συστάσεις του ΕΣΠΕΛ. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαλαβράκος. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, παρότι εν με κάλυψαν οι απόψεις της Επιτροπής, Θέλω να πω ότι ε, διότι και από τη μια πλευρά πρέπει να υποθάλπουμε την προσφυγή στην ε, Επιτροπή μας των διαφόρων πολιτών της Ευρώπης, από την άλλη να τους δίνουμε και ορισμένε οδηγίες ώστε αυτές οι προσφυγές να είναι πιο σωστά διατυπωμένες. Βλέπω ότι μιλάμε για εικαζωμένη κατάχρηση χρηματοδοτικών πόρων. Οι εικαζομένοι αυτοί η οποία βασίζεται στο γεγονός ορισμένων συγγενειών σε σχέση με του αυτούς οι οποίοι ενέκριναν και ανέλαβαν το έργο δεν έχει βεβαιωθεί διαδικαστικής αποφάσεως και αισθάνομαι την ανάγκη ε, να πω ότι θα ήθελα και προσωπικώς να ενημερωθώ από το θέμα, επί του θέματος διότι δεν πρέπει παραβάσεις της ελληνικής ποινική νομοθεσίας να μένουν χωρίς τιμωρία. Το δεύτερο το οποίο έχω να πω είναι ότι δεν θα συμφωνήσω με τον εκπρόσωπο του αναφέροντος ο οποίος είπε ότι στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα κύριε. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι είναι ανέντιμοι που στατιστικά υπάρχει σε όλα τα κράτη αυτή η μερίδα των αντίμων ανθρώπων που συμμερίζονται και συμπεριφέρονται με ανέντιμο τρόπο. Δεν θα δεχόμουν αυτή τη γενίκευση επομένως και δεν θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι ο χώρος της αναντιμότητας. Είναι ο χώρος της αναντιμότητας όταν βλέπουμε μια διαφθορά και σε τοπικό επίπεδο διότι εδώ ξεφεύγει από, την, από τον καταλογισμό κάποιες ευθύνη σε μια διαφθορά πολιτικών. Βλέπω σε ένα τοπικό επίπεδο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ποινικώ ελεγκταίοι έκαναν κάτι που κατά την αποψή σας είναι ποινικό κολάσιμο. Αυτούς να τους δούμε. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε όμως και να προσβάλλουμε μια χώρα. Εν πάση περιπτώσει θα έλεγα να μείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή, να δοθούν όλες οι ε, εκκρεμούσες ακόμη επεξηγήσεις και προσωπικά δηλώνω ότι είμαι διαθέσιμος να το ψάξω και, προ, και ως ε, άτομο, ε, ευρωβουλευτής το θέμα για να προχωρήσουμε στον καταλογισμό ορισμένων ευθυνών. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργεί γενικέσεις εναντίον της χώρας οι οποίες εμφανίζονται τόσο ρηχά ενώπιον αυτής της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στον κύριο Σαλαβράκο να συμφωνήσω με τις γενικές διατυπιστώσεις του που αφορούν ε, στην εικόνα που ενδεχομένως διαμορφώθηκε από τις γενικεύσεις του κυρίου ε, του, του αναφέροντος. Ε, να ρωτήσω προηγουμένω την κυρία Ζορμπαλάν είναι εδώ μήπω θα ήθελε να παρέμβει από μεριά τη Επιτροπή για το ζήτημα που αφορά την ουσία του θέματο. Είστε σημειωμένοι εδώ στην κατάστασή μα. Είστε σημειωμένοι ω ναι. ε, παρουσία από μεριά τη Κομισιόν. Σα ευχαριστώ, αλλά με κάλυψε πλήρω ο συνάδελφό μου, ο κύριο Περουλάκη, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ο, ε, ο αναφέρον θα ήθελε να ένα λεπτό να πω το εξή. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σαλαβράκο. Εγώ δεν είπα ότι όλη η χώρα είναι έτσι. Για το όνομα του Θεού και συμφωνώ και με εσά, ε, κυρία Πρόεδρε, ότι είπα λοιπόν ότι για τη χώρα μου, για την δράμα, για αυτού του ανθρώπου και η αναφορά μου, κύριε Σαλαβράκο, είναι μόνο σε αυτού του ανθρώπου. Και... Να, να του ελέγξουμε. Βεβαίω, βεβαίω. Λοιπόν, ε, ε, Επομένω λοιπόν ανακαλώ και λέω ότι δεν είναι όλη η χώρα έτσι, σαφώ και δεν είναι όλη η χώρα έτσι, σαφώ και δεν είμαστε όλοι σε αυτή τη λογική. Όμω εδώ για το συγκεκριμένο που ήρθαμε να συζητήσουμε είναι αυτό. Όσον αφορά να πω, αν μου επιτρέπετε και κάτι στον κύριο Περουλάκη, σαφώ και δεν. Μου επιτρέπετε σαφώς και δεν ε, προκύπτει ότι υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ της Επιτροπής της Ανάθεσης κτλ. Όταν όμως ο προϊστάμενος, είναι το ερώτημα, μιας Επιτροπής, καθότι και δημοσιογράφος μπορώ να ρωτάω, όταν λοιπόν ο προϊστάμενος μιας Επιτροπής δια των οργάνων του ε, δίνει εντολή να γίνει έλεγχος ή, εν πάση περιπτώσει, να οριστούν, ε, αν θέλετε, επιτροπέ προσωρινή παραλαβή ή οριστική παραλαβή. Όταν λοιπόν αυτή η επιτροπή, η οποία πρέπει να στείλει τι τεχνικέ αναφορέ του ΕΣΠΕΛ, πρέπει να τι στείλει στο, των ε, ελεκτή δημοσίων έργων. Δεν το κάνει. Όταν λοιπόν αυτή η Επιτροπή πρέπει να αναφέρει στη διαχειριστική αρχή τη χώρα μου και η διαχειριστική αρχή δεν παίρνει θέση. Όταν λοιπόν αυτή η Επιτροπή δεν έχει κάνει ένα σωρό πράγματα, γιατί εγώ να είμαι καλοπροαίρετο που θέλω να είμαι σε αυτή την περίπτωση και να μην πιστέψω ότι επειδή προϊστάμενο είναι ο άλλο, δίνει κάποια εν πάση περιπτώσει ε, εντολή αν θέλετε, για ποιο λόγο ο υπάλληλο να υπακούσει απόλυτα. Και μην μου πείτε τώρα και με συγχωρείτε για το χαρακτηρισμό ότι ζούμε σε κοινωνία αγγέλων. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλοι όπω το λέτε και έχει δίκιο και ο Σαλαβράκο και η κυρία Πρόεδρο, αλλά από εκεί και πέρα δεν το κατάλαβα γιατί θα πρέπει όλοι δηλαδή να είναι. Γιατί δεν τα κάνανε αυτά, γιατί δεν τα έκανε αυτά η Τεχνική Επιτροπή που ανέλαβε να, να υποπτεύσει το έργο. Για ποιο λόγο. Μπορείτε ε, να ολοκληρώσετε. Τέλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε κύριε Περβλάκη να προσθέσετε κάτι. Θα ήθελα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να πω πάρα πολλά. Απλώ μόνο ότι όπω είπα και πριν υπάρχει αρχή τη επικουρικότητα. Αυτή η υποχρέωση του ελέγχου έχει επιμεριστεί μεταξύ τη Επιτροπή και των Εθνικών Αρχών. Δεν υπάρχει μόνο κάποιο συγγενή ο οποίο αναθέτει σε ένα άλλο συγγενή τον ένα έργο και είναι ο μόνο ο οποίο ελέγχει την εκτέλεσή του. Είναι λάθο το ότι η διαχειριστική αρχή του προγράμματο δεν ενημερώθηκε και δεν προέβησε καμία ενέργεια γιατί η διαχειριστική αρχή του προγράμματος διατηρεί το έργο στην κατηγορία 2 και ως εκ τούτου είναι αδύνατον η τελική αποπληρωμή του. Και αν δεν υπάρξει η επανακατηγοριοποίησή του, δεν μπορεί να γίνει τίποτα περαιτέρω σε αυτό το έργο. Οπότε δηλαδή ήδη υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες του συστήματος οι οποίες ελέγχουν πιθανές παρενέργειες. Ευχαριστώ. Ε, εγώ να ευχαριστήσω. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε να μας ενημερώνετε για τις επόμενες κινήσεις ελπίζοντας ότι η ελληνική πολιτεία η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη το γνωρίζετε καλύτερα αυτά τα χρόνια με τέτοιου είδους φαινόμενα ε, θα αναλάβει τις ευθύνες της και θα συμβαστεί με τις ε, υποδείξεις της ΕΣΠΕΛ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Σημείο 14. Η γνωμοδότηση επί της ανακοίνωσης σχετικά με την 27η έκθεση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου 2009. Η κυρία Άουκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, στα δανέζικα για να γυμναστούν λίγο και οι διερμηνείς, λέει η κυρία Άουκεν. Βέβαια καταλαβαίνετε είναι πολύ εύκολο να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη όσον αφορά το κείμενο της γραμματείας. Το έλαβα όμω τόσο αργά που δεν μπόρεσα να προσθέσω αυτά που θεωρούσα αναγκαία να προσθεθούν ούτω ώστε να σχηματίσετε πλήρη εικόνα, όμως είναι μια έξοχη επισκόπηση των όσων συμβαίνουν, ποιες διαδικασίες επίσημες ε, υπάρχουν και εφαρμόζονται και θεωρώ ότι όλα αυτά βοηθούν πολύ. Το επόμενο βήμα όμως θα πρέπει να τονίζονται συγκεκριμένα ζητήματα που μας επηρεάζουν εμάς και μας αφορούν εμάς στη δική μας την Επιτροπή και επηρεάζουν και τους πολίτες που στρέφονται προς την Επιτροπή μας. Θα πρέπει επίσης να δούμε ποιο είναι το πρακτικό, ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Θέλουμε να στείλουμε τα μηνύματα στην Νομική Επιτροπή αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, ούτω ώστε να δουν τι πιστεύουμε ότι λειτουργεί και τι πιστεύουμε ότι δεν λειτουργεί. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να προτείνουμε στην Νομική Επιτροπή που έχει, να δημιουργήσει ομάδα εργασίας που θα θεσπίσει εναρμονισμένους κανόνες για την καλή, την ορθή διοίκηση. Αυτό είναι κάτι που ισχύει σε ό,τι κάνουμε. Η σωστή διοίκηση και διαχείριση. Όταν πηγαίνει ο διαμεσολαβητής, ο συνήγορο του πολίτη, όπω πηγαίνει στα διάφορα κάτι μέλη, και αυτά που κάνουμε εμείς, όλα αυτά εμπίπτουν στην σωστή, στην καλή διακυβέρνηση, στην σωστή διοίκηση. Αυτό χρειάζονται οι πολίτες. Χρειάζονται μια σωστή, μια καλή διοίκηση. και πρέπει να είμαστε σαφέστεροι όσον αφορά τα μηνύματα που στέλνουμε στη Νομική Επιτροπή και θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Θέλουμε κανόνες αφέστατους. εύληπτους, εύκολο να εφαρμοστούν. Θα ήθελα να επιστρέψω στο θέμα του νομικού κόστους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και αυτό είναι μια πτυχή της σωστής ε, διακυβέρνησης, της σωστής διοίκησης. διότι αν είναι δύσκολο να προσφύγει κανείς στο δικαστήριο, αν κοστίζει πολύ να προσφύγει κανείς σε ένα δικαστήριο, τότε δεν μπορούν να απολαύσουν τα δικαιώματά του οι πολίτε. Και δεν μπορούν να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι οι νόμοι του κράτους εφηγραμμίζονται πλήρως με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και ήθελα να πω ότι η πρόθεσή μου είναι να προσθέσω αυτά τα στοιχεία το ταχύτερο δυνατόν ούτως ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε το ζήτημα στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας τον Απρίλιο. Ε, έχουμε ειδοποιηθεί για το χρονοδιάγραμμα της Νομικής Επιτροπής. Η έκθεσή τους θα υποβληθεί τον Ιούνιο, άρα χρειαζόμαστε ένα σχέδιο κειμένου τον Απρίλιο. Χρειαζόμαστε και χρόνο για τη συζήτηση επί του κειμένου, για την υποβολή τροπολογιών, ούτως ώστε να στείλουμε τα έγγραφα αυτά στη Νομική Επιτροπή και μπορούμε να αναμένουμε η έκθεση να υποβληθεί στην Ολομέλεια προς έγκριση τον Ιούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και συνάδελφοι. Αυτή ήταν η γενική επισκόπηση των όσων συμβαίνουν και με τα χαράς να ακούσω ποια είναι τα σχόλιά σα επί του θέματο και οδήποτε πληροφορία θα ήταν πρόσδεκτη ούτως ώστε να έχω κάποιε πληροφορίε να εντάξω στι εργασίε μου. Ευχαριστώ κυρία Ούκεν για τι εργασίε σα. Ρωτώ τους συναδέλφους αν θέλουν να τοποθετηθούν. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είναι εδώ. Ο κύριος κρόγκερ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προφανώς σε αυτή τη φάση είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε την εισηγήτρια με κάθε τρόπο. Θα έρθω να σας δώσω την κάρτα μου για να ε, έχουμε την συνεισφορά που ζήτησε η κυρία Βουλευτής. Va bene, eh, Η μόνη μου προσθήκη να ζητήσω από τις διάφορες αντιπροσωπείες να μου δώσουν τα ονόματα των σκιωδών εισηγητών. κυρία... Εντάξει κυρία Μπασέσκου, αλλά λείπουν οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις. Τελειώνει η συνεδρία της Επιτροπής μας και ξεκινάει η συνεδρίαση των συντονιστών.